Καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί έχουμε να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Προβλέπετε ότι η Επιτροπή μας για το θέμα αυτό μέσω του συναδέλφου Beauty Coffer θα κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα των ε, πρώτων υλών. Το θέμα των πρώτων υλών είναι ένα κεντρικό θέμα για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και γι' αυτό, όπως είχαμε υποσχεθεί, ξεκινάμε νωρίς μέσα στη χρονιά με μια ακρόαση με εξαιρετικά σημαντικούς προσκεκλημένους. Καλωσορίζω όλους τους προσκεκλημένους και παραλαμβάνω το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι κατανοούν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και ε, περιμένουμε ακόμη την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής. Υπάρχουν συνεχώς αλλαγές της νομικής βάσης ε, και δεν έχει γίνει δυστυχώς καμία πρόοδος, πράγμα που δεν μας διευκολύνει τη συνέχιση των εργασιών μας πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε και να περιμένουμε ε, την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, και σιγά σιγά να ε, προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή πολιτική γραμμή. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ακόμη τα υποστηρικτικά έγγραφα της Επιτροπής, αλλά θα περιμένουμε. Καλωσορίζω τους προσκεκλημένους μας ίσως ε, να έχουν καθυστερήσει κάποιοι να μην κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας καταρχήν το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπιούτι Κόφερ, για να κάνει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Για την ακρόαση αυτή επιλέξαμε το θέμα μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. για την βιομηχανία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της τροφοδοσίας με πρώτες ύλες. Είναι μια κοινή διαπίστωση και η πολιτική για τις πρώτες ύλες ε, είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική του business as usual. Πρέπει να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για να ασχοληθούμε με, του, με τις πρώτες ύλε. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη της βιομηχανίας ε, για τις πρώτες ύλε. Στο παρελθόν δεν ήταν τόσο μεγάλη η πίεση, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ο μετασχηματισμός προς μια οικονομία που θα επιβαρύνει ως το δυνατόν λιγότερο το κλίμα, οι πρώτες ύλε και η αναζήτηση πρώτων υλών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχουν ε, χώρες ε, που είναι ε, πλούσιες σε πρώτες ύλες και που δεν είναι πάντοτε απόλυτα πρόθυμες να είναι οι μόνιμοι προμηθευτές μας και γι' αυτό χρειάζεται μια σωστή στρατηγική για τις πρώτες ύλε και, όχι απλώς να θεωρούμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε πρώτες ύλε όποτε θέλουμε και όπου θέλουμε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των πρώτων υλών και πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Όταν η γενική οικονομική και πολιτική προοπτική κινείται προς την κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ε, και όταν αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε, η αποτελεσματικότητα πρέπει να είναι ένα βασικό μας μέλημα. Δεν μπορούμε ε, βέβαια να μιλάμε για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αν δεν έχουμε καν πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα για τις σπάνιες γεές και τον ε, ε, τελευταίο χρόνο έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία το θέμα αυτό των σπάνιων γιών και βλέπουμε ότι τα προβλήματα στον τομέα των πρώτων υλών οξύνονται. Πρέπει να ακολουθήσουμε αποτελεσματικότητα λοιπόν στη στρατηγική μας ε, και να έχουμε τις σωστές συνεργασίες. Αυτό ισχύει και εσωτερικά στη συνεργασία με, μεταξύ των δημοσίων αρχών. Ε, ισχύει στο ότι πρέπει να φροντίσουμε από οικολογικής πλευράς τα θέματα, αλλά ισχύει και στις διεθνείς μας συνεργασίες και γι' αυτό σήμερα έχουμε και προσκεκλημένους από πολλές χώρες για να εμπλουτίσουμε το φάσμα της εμπειρίας μας. Είναι σημαντική συνεργασία και με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, βιομηχανικέ χώρε που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση με τη δική μα και χώρε που είναι και πλούσιε ε, σε πρώτε ύλε. Και στι 3 Φεβρουαρίου εδώ στο Κοινοβούλιο θα έχουμε προσκεκλημένους από το Τόκιο, από τη βιομηχανία και το εμπόριο καθώς και από τον τομέα των επιχειρήσεων για να διεξαχθεί μια συζήτηση για τη στρατηγική της Ιαπωνίας για τις σπάνιες γέες. Τέλος, θέλουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκή, μια στρατηγική για την Ευρώπη. που είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να έχει μια εταιρική σχέση για το θέμα των ε, πρώτων υλών, αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη που μπλοκάρουν αυτή τη στρατηγική. Η Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία άρχισαν να αναπτύσσουν δική τους στρατηγική για τις πρώτες ύλε και πρέπει να δούμε όλες οι χώρες μαζί ε, ε, τι θα κάνουμε και οι σημερινές μας εργασίες θα συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή του να βρούμε δηλαδή μια αποτελεσματική στρατηγική για τις πρώτες ύλε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Και πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, ε, θα ήθελα να πω για τους συναδέλφους της Επιτροπής, πριν το ξεχάσω, σχετικά με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης που θα ακολουθήσουν, ότι έχουν αλλάξει μεταξύ τους τα σημεία 6 και 9 της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και ξεκινάμε με τον κύριο Στέφαν Τσόμα. που είναι αντιπρόεδρος ε, για κρατικά θέματα στη UMICOL. Έχουμε περιορίσει το χρόνο ομιλία για να δώσουμε σε όλους χρόνο και να έχουμε και χρόνο συζήτησης. Ο κύριος Τσόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Θέλω να εστιάσω την παρέμβασή μου για να δώσω απάντηση σε τέσσερα διαφορετικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι η τωρινή κατάσταση σε σχέση με τους πόρους τους, τις πρώτες ύλες για τη βιομηχανία ανακύκλωσης. Όταν μιλάμε για ανακύκλωση, μιλάμε για πάρα πολλά υλικά, για πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν θα μιλήσω για τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Επίσης υπάρχουν και ορισμένες ουσίες, ορισμένα προϊόντα, τα οποία μπορούν να ανακυκλώνονται στο διηνεκές, κάτι το οποίο τα κάνει πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης η ανακύκλωση μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκή βάση, σε, σε παγκόσμια βάση και δεν είναι απόλυτα ίδια προβληματική, παρά το γεγονό ότι είναι πολύ παρόμοια. Στην ε, Ευρώπη το κύριο πρόβλημα είναι η πρόσβαση σε απόβλητα από τις ε, πόλεις. Έχουμε προβλήματα με τα απόβλητα των οικοκυριών, με τις ε, χώματερές και με την εξαγωγή ορισμένων από αυτά τα απόβλητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πρόβλημα τεχνολογιών, χρησιμοποίηση τεχνολογιών <clears throat> και σε πολλές χώρες δεν υπάρχει η δυνατότητα πολλά από τα υλικά τα οποία βρίσκονται στα ανακυκλούμενα προϊόντα δεν μπορούν να ανακτηθούν και αυτό οδηγεί σε μεγάλη αναποτελεσματικότητα και απώλεια για πάντα ορισμένων υλικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διάφορα υλικά, τα διάφορα μέταλλα καταρχήν, οι διάφορε βιομηχανίε που χρησιμοποιούν αυτά τα μέταλλα έχουν διαφορετικά προβλήματα. Ο χαλκό και το αλουμίνιο, που είναι σημαντικά βασικά προϊόντα, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ε, διότι απαιτείται και ενέργεια για την ανάκτηση αυτών των υλικών. Πολλά απόβλητα τα οποία έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές εξάγονται παράνομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε πει τις σπάνιες γεές και το λίθιο που δεν ανακυκλώνονται για λόγους τους οποίους, στους οποίους θα επανέλθω. Γιατί λοιπόν έχουμε την ανακύκλωση, έχουμε την ανακύκλωση γιατί υπάρχει κάποια υπολοιπόμενη αξία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η αγορά. Επίσης γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο όγκος αυτών των αποβλήτων ή, <clears throat> ή επειδή υπάρχουν κάποια χρήσιμα υλικά τα οποία βρίσκονται στα προϊόντα τα οποία είναι απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη η σπάνιση αυτών των υλικών και πολλές φορές ακόμα και αυτά τα οποία δεν είναι οικονομικά βιώσιμο να τα ανακυκλώσουμε. Επειδή είναι σπάνια υλικά, στο μέλλον μπορεί να αναγκαστούμε να τα ανακυκλώσουμε. Και αυτό είναι μια σημαντική οπτική γωνία μέσα στα πλαίσια τη αντιμετώπιση ανακύκλωση. Αναξάρτητα όμω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανακύκλωση στην Ευρώπη, είτε αν δεν μπορεί να επιτύχει την κατάλληλη ικανότητα ανακύκλωσης ή αν δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τις περισσότερες επενδύσεις που χρειάζεται, Σίγουρα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη συλλογή υλικών και ανακύκλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για την βελτίωση τη ανακύκλωσης και την επέκτασή της, κάτι το οποίο θα σημάνει και μείωση τη εξάρτηση από εισαγόμενε πρώτε ύλε. Σημαίνει επίσης ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, δυνατότητα επενδύσεων, ευκαιρίε θέσεων απασχόληση, μεγιστοποίηση τη ανάκτηση πρώτων υλών και με την καλύτερη τεχνολογία που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη μπορούμε να συμβάλλουμε και στη μείωση της, του αντικτύπου στην κλιματική αλλαγή, διότι η ανακύκλωση είναι πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων. Το ερώτημα είναι τι ρόλο μπορεί να παίξει η βιομηχανία ανακύκλωση για να εξασφαλίσει η ασφάλεια πρώτων υλών. Πρέπει να σας υπενθυμίσω καταρχήν τι ακριβώς σημαίνει ανακύκλωση μερικοί θεωρούν ότι είναι απλώς η συλλογή υλικών και κάποια ε, διάλυση προϊόντων. Όχι, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα με μια σειρά από βήματα. Φυσικά αν δεν υπάρξει συλλογή δεν μπορεί να υπάρξει ένα κύκλος. Είναι πάρα πολύ η συλλογή των προϊόντων, η διάλυση των προϊόντων τα οποία έχουν συλλεγεί, η πρώτη επεξεργασία και τελικά η ανακύκλωση και ο εξευγενισμός των υλικών που περιέχονται στα προϊόντα αυτά. Μόνο όταν γίνονται αυτά, μόνο όταν έχουμε ανακτήσει τις αρχικές βασικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέα προϊόντα, τότε έχει κλείσει ο βρόχος ανακύκλωσης. <clears throat> Τι μπορεί να κάνει τώρα ο τομέας ανακύκλωσης. Μπορεί να μεγιστοποιήσει το... την έκταση αυτού του βρόχου. Να σας δώσω ε, μερικά παραδείγματα. Τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές περιέχουν υλικά που είναι το ισοδύναμο της πρωτογενούς παραγωγής ως εξής. 600 τόνοι άργυρου είναι 3% της παγκόσμιας παραγωγής. 4% του χρυσού 100, 100 τόνοι, 35 τόνοι παλαδίου είναι 52% της παγκόσμιας παραγωγής, 14.000 τόνοι κοβαλτίου είναι 40, 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές είναι εύκολο να συλλέγονται και να χρησιμοποιείται η καλύτερη τεχνολογία για την ανακύκλωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι το 1 πέμπτο του κοβαλτίου που εξορίσετε σήμερα θα μπορούσε ήδη να αποκτάται από την ανακύκλωση. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει την συγκέντρωση αυτών των προϊόντων που βρίσκονται σε ε, ανακύκλωση. Σε ένα τόνο ε, ορυκτού έχετε 5 γραμμάρια χρυσού. Αλλά σε ένα τόνο ε, πλακετών υπολογιστή έχετε 200 γραμμάρια. Και σε ένα τόνο κινητών τηλεφώνων έχει 20 με 30 γραμμάρια για τις άλλες ουσίες οι οποίες είναι ευγενή μέταλλα, ρόδιο, παλάδιο, πλατ, ε, πλατίνα, έχετε 2 κιλά αυτών των υλικών και όχι 5 γραμμάρια μονάχα στα, στο πρωτογενές ορυκτό. Επομένως, όλα αυτά τα απόβλητα που βγαίνουν από αστικές περιοχές είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πλούσια σε πρώτες ύλες και αν μπορούμε να τα συλλέξουμε όλα αυτά και να τα ε, να εξαγάγουμε αυτές τις ουσίες είναι πολύ θετικό για την βιομηχανία. Για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση στη βιομηχανία χρειαζόμαστε υψηλή τεχνολογία, μεγάλες επενδύσεις και φυσικά οικονομία κλίμακος. Και η ευρωπαϊκή βιομηχανία ανακύκλωση αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κάνει περισσότερες επενδύσεις για να ξεπεράσει μια σειρά από προσκόμματα και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Τέταρτον, χρειάζεται καινοτομία. Μπορούμε πάντα να καινοτομούμε για να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης για νέα προϊόντα τα οποία έρχονται στην αγορά. Για να κλείσω το δεύτερο ερώτημα, μπορεί να κάνει τη διαφορά ο τομέας της ανακύκλωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των, ε, για τις πρώτες ύλες και την αποτελεσματική χρήση τους, γιατί μπορεί να μας δώσει αυτές τις ουσίες οι οποίες είναι σπάνιες, Εάν υπάρξει σωστή συλλογή, σωστή διάλυση των ε, προϊόντων, εάν δεν εξάγονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι παράνομος και αν τυχάνουν επεξεργασίας και εξευγενισμού με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Πού είναι τώρα τα εμπόδια, ιδίως για τις κρίσιμες πρώτες ύλε. Σας υπενθυμίζω ποιες είναι αυτές οι ουσίες. Σήμερα είναι τα μη σιδηρούχα μέταλλα. Τα κρίσιμα αυτά ε, υλικά χρησιμοποιούνται σε πολύπλοκες ε, ε, εφαρμογές. Έλεγχος εκπομπών, ανανεώσιμη ενέργεια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Όσο πιο πολύπλοκη είναι η εφαρμογή στην οποία χρησιμοποιούνται, τόσο πιο πολύπλοκη είναι και η διαδικασία ανακύκλωσης και τα διάφορα βήματα στην αλυσίδα ανακύκλωσης και η τελική διαδικασία εξευγενισμού. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανακύκλωσης εξαρτάται φυσικά από την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα κάθε ενός από τα βήματα στην αλυσίδα. Ο πιο αδύναμος κρίκος είναι το βήμα αυτό το οποίο έχει τη χαμηλότερη αποδοτικότητα και αυτό καθορίζει τη συνολική αποδοτικότητα της όλης διαδικασίας. Ένα <coughs> χαρακτηριστικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και ξαναγυρίζω στην αλυσίδα ανακύκλωσης είναι η συλλογή. Ένα παράδειγμα το οποίο μου αρέσει να χρησιμοποιώ γιατί είναι πολύ εύκολο να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Μόνο 2% των κινητών τηλεφώνων συλλέγονται και ανακυκλώνονται σήμερα. 2%. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η ανεπαρκής διάλυση. Σε ένα αυτοκίνητο που φτάνει στο τέλος της ζωής του, Εάν δεν φύγουν τα ηλεκτρονικά από ένα αυτοκίνητο προτού πάει στην πρέσα, τότε χάνονται τα μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία βρίσκονται στα ηλεκτρονικά του αυτοκίνητου. Πρέπει λοιπόν προηγουμένω να αποσύρονται, να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο. Ένα άλλο παράδειγμα, άμα πάρετε ένα κινητό τηλέφωνο και αρχίσετε να το διαλύετε, να το κάνετε φύλλο και φτερό, ορισμένα πολύτιμα μέταλλα θα φύγουν μαζί με το πλαστικό. Και σε αυτή την περίπτωση θα χαθούν. Πρέπει απλώς να βγάζει κανείς την μπαταρία από το κινητό τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι παραδείγματα λοιπόν που δείχνουν ότι η σωστή διαδικασία διάλυσης εξαρτάται από το είδος του προϊόντος. Επίσης έχουμε κακή διαχείριση <coughs> της ροής που ακολουθεί την πρώτη επεξεργασία. Ιδίως όταν μιλάμε για κρίσιμα, σπάνια υλικά τα οποία εμφανίζονται ως ίχνη μονάχα στα διάφορα προϊόντα, αν δεν υπάρχει σωστή διαδικασία ανακύκλωσης και καταλήξουν σε μια συνολική διαδικασία, είτε πρόκειται για χάλιβα είτε για αλουμίνιο, θα χαθούν τα σπάνια υλικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία και δεν υπάρχει δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν. Τέταρτον, η σωστή ανάκτηση και εξευγενισμός των υλικών. Όταν μίλησα για την παράνομη εξαγωγή προϊόντων, τα υλικά αυτά που πηγαίνουν σε αναδυόμενες χώρες όπου δεν υπάρχει απόλυτα η απαραίτητη τεχνολογία, πολύ συχνά τουλάχιστον, περίπου 25% του χρυσού που βρίσκεται στις, ε, στα προϊόντα αυτά ανακτάται και μόνο το χρυσάφι ανακτάται, ενώ η καλύτερη τεχνολογία μας επιτρέπει σε άλλες χώρες να έχουμε το 100% του χρυσού και πολλά άλλα, καμιά εικοσαριά άλλα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και για την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο. Γιατί αυτά τα υλικά χάνονται για πάντα. Τέλος, η επαναχρησιμοποίηση, αντικατάσταση ή ανακύκλωση συνήθως μπορούν να γίνουν και τα τρία. Η αναχρησιμοποίηση είναι η καλύτερη λύση εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητε προποθέσει. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η ανακύκλωση στο τέλο ζωή ενό προϊόντου. Παραδείγματο χάρη, ένα κινητό τηλέφωνο το χρησιμοποιήσετε σε τρία χρόνια και να το πετάξετε σε μία χωματερή, είναι χειρότερο από το να το ανακυκλώσετε μετά από ένα χρόνο μονάχα, γιατί μπορεί να ανακτηθεί το υλικό του και ξαναχρησιμοποιηθεί. Επομένω, η επέκταση τη ζωή ενό προϊόντο θα πρέπει να γίνεται μονάχα αν μπορεί να ανακυκλωθεί στο τέλο. Και επίση θα πρέπει να προτιμούμε να υπάρχει πλήρη ανακύκλωση. Αν μας ενδιαφέρει μόνο να ανακυκλώσουμε ένα κομμάτι του εξοπλισμού, αυτό να το παραχρησιμοποιήσουμε, αυτό έχει νόημα μονάχα αν το υπόλοιπο θα ανακυκλωθεί. Μπορείτε να παραχρησιμοποιήσετε το τσίπ με του κινητού τηλέφωνου, αλλά μόνο αν δεν σταλούν τα άλλα στη Πολλές φορές υπάρχει η ψευδής δήλωση επαναχρησιμοποίησης ή οι παράνομες ε, εξαγωγές. Η αντικατάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδέα όταν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ορισμένε κέρυες ύλες όπως είναι μέταλλα και ε, υφαντουργικά και όταν τα υλικά υποκατάστασης μπορούν και αυτά να τύχουν στη συνέχεια ανακύκλωσης. Θέλω να κλείσω λοιπόν στο σημείο αυτό ότι για να εξασφαλίσουμε μια αποδοτική καλύτερη τεχνολογία Χρειάζεται καλή συλλογή και εδραίωση της διαδικασίας συλλογής, καλές διαδικασίες διάλυσης και πρώτης επεξεργασίας. Όλα αυτά πρέπει να εξασφαλιστούν. Πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες εξαγωγές. Και αυτό ισχύει για την Ευρώπη, αλλά ισχύει και για το υπόλοιπο τμήμα του κόσμου, όπου υπάρχει πραγματική θέληση να βελτιωθεί η ανακύκλωση. Το τέταρτο ερώτημα τελικά, τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και οι άλλοι εμπλεκόμενοι για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωση και επομένω η ασφάλεια των σπανιών πόρων. Οι κυβερνήσει πιστεύουμε ότι πρώτα πρέπει να εφαρμόσουν με ενιαίο τρόπο και να ελέγξουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί υπάρχει καλή νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πλήρης και ενιαίος και δεν υπάρχει απόλυτη αστυνόμευση παραγωγός χάρη η υγιής διαχείριση για τα θέματα του περιβάλλοντο και η απαγόρευση των εξαγωγών είναι ένα παράδειγμα και η ανεπαρκή συλλογή υλικών σε πολλά είναι ένα άλλο παράδειγμα. Χρειαζόμαστε τα πρακτικά μέσα για να εξασφαλίσουμε αυτόν τον έλεγχο τη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ένα πρόβλημα είναι το θέμα του ελέγχου των εξαγωγών από την Ευρώπη. Πρέπει να βρούμε εργαλεία τα οποία είναι αποτελεσματικά για τον έλεγχο αυτό. Είναι απαραίτητη η αποτελεσματικότητα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να προωθήσουμε την συλλογή υλικών στο τέλος της ζωής τους. Και πρέπει η ανακύκλωση να αντιμετωπίζεται συστημικά, σαν σύνολο. Γιατί πολλές φορές δίνουμε έμφαση σε ένα μονάχα κομμάτι της αλυσίδας και όχι τα υπόλοιπα. Αν δούμε μονάχα ένα κομμάτι της αλυσίδας, αυτό το κομμάτι μπορεί να ενισχυθεί, αλλά θα είναι σε βάρος της σύνολης αλυσίδα. Αν μα απασχολεί μονάχα η συλλογή. Θα πάρουμε υλικά, θα τα συλλέγουμε, θα τα διαλύουμε και θα τα εξάγουμε. Αυτό δεν θα οδηγήσει τίποτα στην Ευρώπη. Δεν θα έχουμε πραγματική ανάκτηση υλικών παρά την καλή συλλογή. Πρέπει να σκεφτόμαστε ολιστικά, πρέπει να σκεφτόμαστε όλο το βρόχο ανακύκλωση σαν σύνολο. ο συνδυασμός της αποτελεσματικότητας και η ασφάλεια για τους ε, για την ανάκτηση πόρων είναι τμήματα μιας συνολικής λύσης <clears throat> και επίσης θα πρέπει να δώσουμε στο, στην προσπάθεια ανακύκλωσης να δώσουμε έμφαση στις κρίσιμες προτεσίλες οι οποίες δεν ε, υπάρχουν σε μαζικό επίπεδο. Μας νοιάζει μονάχα ο όγκος ανακύκλωσης. Ξεχνάμε το να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν μερικά κρίσιμα υλικά τα οποία πρέπει να ανακτηθούν. Ποιότητα λοιπόν στην ανακύκλωση και όχι μονάχα ποσότητα. Και για τον βιομηχανικό τομέα θα πρέπει να λειτουργήσουμε για μια αλυσίδα παραγωγής αξίας και όχι μονάχα σε ένα κλειστό κύκλο ο οποίος αφορά μονάχα τη βιομηχανία και τους ανακυκλωτές. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να καινοτομούμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις οι οποίες έρχονται από τις νέες τεχνολογίες και τα νέα προϊόντα που έρχονται στην αγορά πρέπει να επενδύσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα, να έχουμε μια κυκλική χρήση των προϊόντων και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά λοιπόν, εάν αντιμετωπιστούν και επιληθούν, θα μας δώσουν τις απαραίτητες ποσότητες οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Τέλος, οι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις κτλ. θα πρέπει να προωθήσουν την προσέγγιση με αλυσίδα προσθέμενης αξίας, να προωθήσουν την κυκλική αντιμετώπιση των προϊόντων και μια ολιστική προσέγγιση η οποία συμπεριλαμβάνει και τους καταναλωτές και τους ερευνητές και τους άλλους εμπλεκόμενους. Οι διεθνείς φορείς και οι οργανισμοί θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο επίση και νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουν περιφερειακές πρωτοβουλίες για να επιταχυθεί η σύνολη διαδικασία. Να έχουμε ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Εν κατακλείδη λοιπόν είναι καιρό να κάνουμε κάποιε θεμελιώδει αλλαγέ και να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα για να ξεπεράσουμε την ιδέα τη διαχείριση αποβλήτων και να περάσουμε στη διαχείριση πόρων. Να μην κοιτάζουμε μονάχα τον όγκο, αλλά τον όγκο και την ποιότητα από την αντιμετώπιση αποβλήτων σε ανακύκλωση ε, προϊόντων υψηλή αξία. Δεν είναι μια εύκολη ιδέα στο τέλο τη ζωή ενό προϊόντο να το ανακυκλώσουμε. Είναι διαδικασία που μπορεί να δώσει μεγάλη αξία. Και τέλος, η βιομηχανία θα πρέπει να δει την ανακύκλωση όχι σαν άχθος, αλλά σαν ευκαιρία. Αν υπάρχει λοιπόν νομοθεσία η οποία έχει βοηθήσει την κατάσταση στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος για τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, αυτό οδηγεί σε μεγάλη διαφορά μεταξύ Ευρώπης και άλλων χωρών του κόσμου. Η σωστή αντιμετώπιση για τους σπάνιους πόρους λοιπόν είναι απαραίτητη. Το να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μία εξασφάλιση της ε, διατήρησης των πόρων αυτών και του να έχουμε μια κυκλική οικονομία για τα προϊόντα αυτά. Αυτά μπορεί να γίνει με την κατάλληλη νομοθεσία και εφαρμογή. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσόμα. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στεφάν Αχντητή. είναι υπεύθυνο ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο ε, για θέματα προϊόντων και αποβλήτων. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Morning, everybody. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια κρύωση για την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες και τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο είναι μια ομοσπονδία εθνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων Απλώς ενημερωτικά σας το λέω. Έχουμε κάποιες διαφάνειες, νομίζω ότι μπορείτε να τις δείτε. Ελπίζω να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποια ερωτηματικά, τα οποία θα διευκρινιστούν ε, μέσω συζήτησης. Στην παρέμβασή μου θα εστιάσω σε δύο σημεία κυρίως. Το πρώτο είναι η ασφάλεια των πόρων και ορισμένες φορές δημιουργούνται νέες ε, δυνατότητες και αμφισβητείται ο τρέχον τρόπος ζωής μας. Βλέπετε το διάγραμμα εδώ και έχετε τις τάσεις για τις βασικές ε, ε, καταναλώσεις πόρων που κάνουμε. Όπως διαπιστώνετε, στα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιούμε ακόμα και περισσότερα, ε, περισσότερους φυσικούς πόρους και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα 30 χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν είναι μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι ή όχι. Και νομίζω ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλε θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της ε, κατανάλωσης ε, των ε, πόρων μας και του πώς, πώς τους διαχειριζόμαστε. Η δεύτερη διαφάνεια είναι τεχνικής φύσεως, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσει να χρησιμεύσει για να διευκρινίσουμε και να θέσουμε κάποια θέματα. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στην αποσύνδεση. Λες και πλέον μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερο, ε, περισσότερες οικονομικές αξίες χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον ισχύει αυτό. Δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σε άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος μέτρησης της αποσύνδεσης της ε, κατανάλωσης πόρων σε σχέση με τις οικονομικές αξίες. Το δεύτερο σημείο της παρέμβασής μου και νομίζω ότι εκεί ε, τίθεται και τα περισσότερα ερωτηματικά είναι ε, η εσωτερική κατανάλωση και οι δυνατότητες που έχουμε εμείς εσωτερικά. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά ποια είναι τα πιο χρήσιμα και τα πιο προσβάσιμα υλικά που έχουμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προλαλήσαντα, ο οποίος μας υπονδύμισε τι σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν στην ανακύκλωση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, θα πρέπει να έχουμε αστική ε, συσσόρευση πολυβλήτων ή ε, των γεών. Ε, χρησιμοποιούμε πλέον 16 τόνους ε, από, πόρων και παράγουμε περίπου 3,5 τόνους, συγγνώμη, εισάγουμε περίπου 3,5 τόνους πόρων. Το ερώτημα είναι λοιπόν πού θα πρέπει να δεθεί προτεραιότητα. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την πρωτοβουλία είναι να υπάρχει και το ανάλογο θάρρος να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιους πυλώνες. Υπάρχουν τρεις πυλώνες σε αυτή την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε. Νομίζω ότι τους γνωρίζετε παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί το τελευταίο έγγραφο. Και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ο τρίτος πυλώνας. Δηλαδή να ασχοληθούμε πρώτον με το θέμα της κατανάλωσης πόρων και πώς μπορούμε να έχουμε αποδοτικότητα των πόρων, ε, να δώσουμε μια νέα όθηση στην ανακύκλωση πριν εξετάσουμε νέες στρατηγικές ε, για τα θέματα της εξόρισης γεών και ε, του διεθνούς εμπορίου μην θεωρήσετε ότι ε, πιστεύω ότι είναι άχρηστα όλα τα μέσα που έχουμε στους άλλους πυλώνες. Ε, σε καμία περίπτωση, απλώς θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτή η προτεραιότητα. Από αυτά που θα μπορέσουμε να έχουμε από τον ε, πρώτο πυλώνα, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για το δεύτερο και τρίτο πυλώνα. μου ζητήθηκε επίσης να απαντήσω και ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για τα αποτελέσματα της εξόριξης γεών για τη βιοπικιλότητα. Αυτό που έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση είναι να θα σα υπενθυμίσω το εξή. Παρά το γεγονό ότι είναι δύσκολο να μετρήσουμε τη βιοπικιλότητα αυτή τη στιγμή, ε, είναι ίσως η μεγαλύτερη μας ανησυχία. Όταν λοιπόν ασχολούμαστε με την εσωτερική εξόριξη, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι αυτό που χρειαζόμαστε και αν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για μας. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, έχετε και τα πιο σημαντικά στοιχεία. Αν δούμε τον κατάλογο των ε, βασικών υλικών τα οποία ε, έχει ε, επισημάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι δημόσια, βλέπετε ότι όλα τα σπάνια και πολύ κρίσιμα υλικά δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο σημαντικά. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Χρειάζεται τώρα ως πρώτο βήμα να έχουμε πιο έντονη εσωτερική εξόριξη όταν γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις πιο σημαντικές πρώτες ύλες όπως μας υπενθύμησε και ο Στεφάν είναι σαφώς πολύ πιο συγκεκριμένες, ε, συγκεντρωμένες στα αστικά μας απόβλητα παρά στα περισσότερα ορυχεία, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει αυτό λοιπόν να το έχουμε κατά νου. Και θα κρατήσω και αυτή τη διαφάνεια εδώ για τα συμπεράσματά μου. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω λίγο περισσότερο στις επιπτώσεις εξόριξης πόρων για τις γέες και τη βιοποικιλότητα. Όσα προληπτικά μέτρα και να λάβουμε για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και αυτό το οποίο αποκαλούμε βιώσιμη εξόριξη πλέον, δεν είναι ε, παρά μόνον έλεγχος των καταστροφών που κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι φυσικό. Υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις για τη γη και τη βιοπικιλότητα σε κάθε εξόριξη. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφώνησε να έχουμε ένα νέο δίκτυο Natura 2000. Και γιατί θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ του Natura 2000 και των εσωτερικών εξορίξεων. Διότι οι εσωτερικές εξορίξεις αφορούν ε, εκτάσεις γης οι οποίες πλέον βρίσκονται στο προστατευόμενο δίκτυο του Natura 2000. Θα πρέπει λοιπόν να αποσταλούν σαφή μηνύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θέλουμε να επεκτείνουμε το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του Natura 2000, δεν θα πρέπει ε, μόνοι μας ε, να ε, αμφισβητούμε τα όσα λέμε και να επιτρέπουμε εξορίξεις σε αυτές τις περιοχές, δεδομένου ότι δεν είναι και αυτό που χρειαζόμαστε, βλέποντας και τη διαφάνεια που σας παρουσίασα. Δεύτερον, τίθεται και το ερώτημα του ποια στρατηγική φέρπει της εσωτερικής ε, εξόριξης. Αν θέλουμε να εξάγουμε περισσότερα ε, σύμπλοκα, μήπως η διάλυση των αποβλήτων θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ. και έτσι δεν θα υποσκάπτουμε και το στόχο της βιοπικιλότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη συζήτηση και όχι να μακρηγορώ εγώ και να συνεχίσω να σας λέω πράγματα στην παρέμβασή μου. Απλώς ένα συμπέρασμα να σας δώσω. Πέραν του τρίτου πυλώνα και της καινοτομίας που ε, θα πρέπει να τον συμπεριλάβουμε και στον τρίτο πυλώνα, οι υπόλοιποι πυλώνες απλώς συνεχίζουν το ίδιο αναπτυξιακό μοντέλο που γνωρίζουμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Κάτι δε που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση είναι ότι ε, οι διεθνείς ε, τάσεις μπορεί να συνεχίσουν να, ε, να εντείνουν περισσότερο τις εντάσεις ε, παγκοσμίως και φοβάμαι ότι δεν θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε καλύτερα τι ωφέλη θα έχουμε αν εντοτικοποιήσουμε τις διεθνείς μας ε, εμπορικές δραστηριότητες και με συγχωρείτε που γίνομαι λίγο προκλητικός, αλλά ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε και κατά πόσον αυτές οι διεθνείς ε, πρακτικές, ε, ε, οι εμπορικές, θα μπορούσαν ίσως να οδηγήσουν σε μια νέα μορφή απεικιοκρατίας. Όπως σας είπα, ο δεύτερος πυλώνας δεν θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι βασικές μας ανάγκες, αλλά θα μπορούσαν ίσως να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα για τους στόχους της βιοποικιλότητάς μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιε είναι οι προτεραιότητές μας στις εσωτερικέ εξερίξει. και νομίζω ότι η σαφή απάντηση είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα την αστική εξόριξη ή την ε, ευρωπαϊκή εφευρητικότητα στα θέματα εξόρυξης. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον τρίτο πυλώνα, να δημιουργήσουμε τις προποθέσει για νέο σχεδιασμό προϊόντων και στρατηγικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα Και στην τελευταία διαφάνεια βλέπετε ότι εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα ε, ψηφίσετε πολύ σημαντικά ε, για κάτι πολύ σημαντικό, συγγνώμη, στις 3 Φεβρουαρίου και πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω να χρησιμοποιήσετε την ψήφο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 3 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ο τελευταίος στο πρώτο αυτό πάνελ είναι ο Δ. Στέφεν Μάιερ ο οποίος είναι μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπιουτικόφερ για την πρόσκληση. Αξιότιμοι κύριε βουλευτές κυρίες βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Λόγω χιονοπτώσεων καθυστέρησα. Ναι, ναι, θα αλλάξω, θα μιλήσω γερμανικά, μην ανησυχείτε. αυτό ήθελα να πω ακριβώ ότι θα μιλήσω γερμανικά γιατί έχω προετοιμάσει την παρουσίασή μου στα γερμανικά. Όπω σα είπα λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ και για την ε, σημασία που αποδίδεται στη στρατηγική των πρώτων υλών και στην ασφάλεια της βιομηχανίας πρώτων υλών. Από το 2008 άρχισε η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει κάνει σημαντικά βήματα. Από την πλευρά της γερμανικής βιομηχανίας πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε να έχουμε φτάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει σήμερα να δημοσιεύσει μία ανακοίνωση για τις πρώτες ύλε ε, και είναι κρίμα που πάλι αναβλήθηκε η ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, χαιρετίζουμε το ότι η δική σα Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα των πρώτων υλών και ετοιμάζει έκθεση για το θέμα των πρώτων υλών και τη στρατηγική στην Ευρώπη. Θα σας πω πώς έχει η κατάσταση στη γερμανική βιομηχανία. Όσον αφορά την ε, ε, προμήθεια πρώτων υλών και σπανίων γεών συγκεκριμένα, ε, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Η Κίνα έχει επιβάλει συγκεκριμένους περιορισμούς και από ό,τι ξέρουμε θέλει να περιορίσει περαιτέρω τις εξαγωγές η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και έτσι η κατάσταση όσον αφορά τις σπάνιες γεές παραμένει προβληματική. Για πρώτες ύλες από άλλες χώρες ε, και πάλι υπάρχουν προβλήματα για τη βιομηχανία. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος και για την, ε, τον εφοδιασμό της βιομηχανίας με πρώτες ύλε, αλλά ε, υπάρχει και ευρύτερο πρόβλημα για τις εμπορικές ροές σε ολόκληρο τον κόσμο. Κυρίως υπάρχουν ε, περιορισμοί από ε, τις εξαγωγές ε, παλιοσίδερων από χώρες όπως η Ρωσία που έχει μειώσει κατά 50% τις εξαγωγές της αλλά και τον τρίτο πυλώνα της, ε, του εφοδιασμού ε, με πρώτες δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση της προμήθειας από ε, τρίτες χώρες. Έχουμε πολύ δύσκολη πρόσβαση σε μερικές φορές και σχεδόν αδύνατη είναι η πρόσβαση στην εξόριξη πρώτων υλών για διάφορους λόγους και προβλήματα υπάρχουν και στον μελλοντικό προγραμματισμό. Η βιομηχανία ασχολείται και με, την, με τους τρεις ε, πυλώνες για την προμήθεια των ε, ε, πρώτων υλών και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και δεν έχει βελτιωθεί. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι βασικό μέλημα της ε, οικονομίας και του κλάδου να μπορέσει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της βιομηχανίας. Τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τις εισαγωγέ πρώτων ε, υλών ε, συμπεριλαμβάνουν τη διαφοροποίηση των προμηθειών και την άμεση συμμετοχή σε εξόριξη πρώτων υλών σε προγράμματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο αυτά εργαλεία μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα η συμμετοχή σε προγράμματα εξόρυξης ε, πρώτων υλών ε, θα μπορούσε να αποτελέσει κάποια λύση. Η Γερμανία εισάγει κάθε χρόνο πρώτες ύλες ε, αξίες πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως μέταλλα. Με άμεση συμμετοχή σε ορυχία και σε εξόρυξη θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτή, αυτός ο εφοδιασμός. θέλουμε να μην υπάρχουν ε, περιορισμοί στο εμπόριο και για μας κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ε, μόνο οι επιχειρήσεις ε, που μπορούν να έχουν αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών και υλικών μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν δυνατότητες επιβίωσης στην παγκόσμια αγορά. Ε, γι' αυτό τονίζουμε το δυναμικό περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην προμήθεια πρώτων υλών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και θα πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστικοί στη συζήτηση με πολύ εμπεριστατωμένα στοιχεία. Προσπαθούμε να έχουμε σαφή στοιχεία για τη χρήση πρώτων υλών, καθώς και τις ε, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικές οι δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρωτεσίλες στην ε, Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα. Ε, ε, θέλουμε να έχουμε και σωστή προστασία σε αυτά τα οποία κάνουμε. Μας ενδιαφέρει και ε, η δευτερογενής προμήθεια πρωτανηλών ε, από άλλες χώρες. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την βελτίωση της βιωσιμότητας και των τριών πυλώνων στον εφοδιασμό πρωτανηλών Μέσω του ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει τον περιορισμό των εξαγωγών από την Κίνα. Οι διαδικασίες του ΠΟΕ είναι μια είναι χρονοβόρες και δεν μπορούμε να περιμένουμε άμεση απάντηση, αλλά με τα μέτρα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της και θα προσπαθήσει να αναπτύξει το διάλογο με τρίτες χώρες με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού ε, επίσης δίνουμε την πρέπουσα σημασία για την ανάκτηση υλικών και δημιουργούνται ε, οι προϋποθέσεις για να μειωθούν οι παράνομες εξαγωγές ε, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Θέλουμε να υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ της σωστής χρήσης ε, ε, των ανακυκλούμενων υλικών και των, ε, της προστασίας των περιοχών στις οποίες μπορούν να διατίθενται τα υλικά αυτά ακόμη μέσω του γενικευμένου συστήματος ε, προτιμήσεων ε, θα γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την πρόσβαση των τρίτων χωρών σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει ε, επίσης και τη σωστή διεξαγωγή συμφωνιών με τρίτες χώρες όπως είναι η Ινδία. Θέλουμε να έχουμε το σωστό πλαίσιο για τις ρυθμίσεις όσον αφορά ε, τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Και θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν καταλήλως ε, οι κατηγορίες ε, ανακυκλούμενων προϊόντων. Ε, τα παλιά αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να εντάσσονται στη σωστή κατηγορία για τα ανακτώμενα υλικά. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν τα σωστά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασκεί το διάλογο με τις χώρες που είναι υπεύθυνε για τις ε, περιοχές του Natura 2000 ώστε να υπάρχει σωστή προστασία ε, του περιβάλλοντος. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να φροντίσει και τα θέματα καινοτομία ε, όσον αφορά την ε, προμήθεια των πρώτων υλών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα και πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Μία σωστή πολιτική εμπορίου που θα αντιμετωπίζει και τις τρευλώσεις ανταγωνισμού, θα χρησιμοποιεί και το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων και κάθε άλλη δυνατότητα. Η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε ε, θα πρέπει να συνεχιστεί και στους τρεις πυλώνες που προανέφερα και να γίνει και σωστά η εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο. δεν είναι προφανές ότι θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες ύλε και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, τάσεις που αναπτύσσονται για το μέλλον. Οι πρώτες ύλε έχουν ε, τεράστια σημασία για την οικονομία μας για το μέλλον και θα βελτιωθούν περαιτέρω οι μελλοντικέ τεχνολογίες χτίζοντας πάνω ε, στα θέματα που αφορούν τις ε, πρώτες ύλε. Ε, θέλουμε να περιορίσουμε το παράνομο εμπόριο σε πρώτες ύλε και να βελτιώσουμε την βάση που έχουμε στην Ευρώπη ώστε να έχουμε μια βιώσιμη στρατηγική. Χωρίς παράλληλα να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη ε, και γι' αυτό θα έχουμε και την κατάλληλη επισήμανση και πιστοποίηση για να βοηθήσουμε τις ε, ευρωπαϊκές ε, εταιρείες. και με βάση την πολιτική της Επιτροπής θα συνδυαστούν τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις προωθώντας την ανταγωνιστικότητά τους και προστατεύοντάς τις από αντίξωες οικονομικές συνθήκες και πτώχευση. Θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων στην Ευρώπη συνολικά και η βελτίωση ε, της βιωσιμότητας είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Η της χρήσης πρώτων υλών από τη βιομηχανία ε, είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ε, των ε, πρώτων υλών και η πολιτική για τις πρώτες ύλε είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του Επιτρόπου κ. Ταγιάννη. Χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία σχετικά με τις πρώτες ύλες και πιστεύουμε ότι θα τύχει και τη σωστή αντιμετώπιση στο θέμα και στην Επιτροπή σας. Η έκθεση αυτή ελπίζουμε ότι θα δώσει την όθηση για τη βελτίωση της χρήσης πρώτων υλών και για την ε, εξασφάλιση των προτύπων της βιομηχανίας για τις πρώτες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που έχουμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων για το πάνελ αυτά και έχουμε τους πρώτους οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο ήδη, ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αγορητές. Το ερώτημα μου είναι πώς ερμηνεύεται την πρωτοβουλία του Ρίτς και τις ε, επιπτώσεις που θα έχει στην ε, απόκτηση <clears throat> πρώτων υλών και την ασφάλεια στην απόκτηση ε, πρώτων υλών. Πώς το αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό το θέμα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι θεωρείτε μέσα στο ότι είναι λογικό μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα να υπάρχει μια κοινή πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά και πώς αντιμετωπίζετε τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες στον τομέα των πρώτων υλών. Θα μαζέψουμε μερικές ερωτήσεις για καλύτερη χρήση του χρόνου. Ο κύριος Μπιτικόφερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θέσω ερωτήματα στον κύριο Τσόμα και στον κύριο Μάια. Κύριε Τσόμα, Είπατε ότι σε ορισμένου τομεί η ανακύκλωση δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο της οικονομικής βιωσιμότητας. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που μπορείτε εσείς να φανταστείτε, να προτείνετε για την ε, πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε για τα σπάνια ή στρατηγικά σημαντικά ε, υλικά τα οποία μπορεί να μην είναι οικονομικά βιώσιμο να γίνει η ανακύκλωσή τους. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, κρίνετε τις προσπάθειες να, ε, να γίνει η ανακύκλωση πιο αποτελεσματική με την ενσωμάτωση της έννοιας της ανακύκλωσης στην οδηγία οικο, οικολογικής σχεδίασης. Δηλαδή ήδη από την αρχή της δημιουργίας ενός προϊόντος να λαμβάνει υπόψη η ανάγκη ανακύκλωσης και προ τον κύριο Μάιο θέλω να θέσω το ερώτημα ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία κατά την άποψή σα είναι απαραίτητα για να καταπολεμηθεί η παράνομη εξαγωγή προϊόντων στην οποία αναφερθήκατε ιδίω για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα ώστε να μειωθεί αυτή η παράνομη εξαγωγή τους. Και ένα ακόμα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω στον κύριο Μάιερ επίσης. Είπατε ήδη πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση για τις πρώτες ε, ύλες από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά και προηγουμένως ο κύριος Αντιτή είπε ότι πολλά από τα στρατηγικά σημαντικά υλικά δεν μπορούν να αποκτηθούν μέσα στην Ευρώπη. Το ερώτημα είναι λοιπόν, κατά την άποψή σας, ποια είναι τα, ποιες είναι οι πρώτες ύλες που πρέπει πράγματι να αναζητηθούν στα αστικά απόβλητα στην Ευρώπη, ποια είναι αυτά που έχουν πραγματικά μεγάλη σημασία και ποιε είναι οι προτεραιότητε που θέλετε να θεσπίσετε σε σχέση με αυτά τα υλικά. Και το τελευταίο ερώτημα. Είπατε πολλές φορές για το περιεχόμενο της πρώτης, του πρώτου σχεδίου ανακοίνωσης της Κομισιόν και την εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Αυτό όμως δεν, δεν εμφανίζεται στο δεύτερο σχέδιο της πρότασης της Κομισιόν. Εγώ δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό, αλλά θεωρείται ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει μια πολιτική έναντι χωρών οι οποίες δεν έχουν, έχουν μεγάλη δυνατότητα να παράγουν ε, πρώτες ύλες με σκοπό να αφαιρέσει από αυτούς την προτιμησιακή ε, εμπορική σχέση όταν δεν, δίνουν εξαγωγή, όταν δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αυτών των προϊόντων. Florence. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και όχι μόνο να τα γενέθλια του κυρίου Μπίτε Κόφερ, είναι σημαντική αυτή η μέρα, αλλά επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση την οποία είχαμε κάνει ήδη πριν από 10 χρόνια ουσιαστικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όταν μιλούσαμε για τα αυτοκίνητα δεν είχαμε τότε τη δυνατότητα για δύο εκθέσεις, την έκθεση 3α και την έκθεση για τα αυτοκίνητα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τέτοιων ρυθμίσεων. Και σήμερα στις 12 η ώρα είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολιών για την οδηγία 3α, η οποία αναφέρθηκε από τον παλιό μας εισηγητή εδώ. Εμείς αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινά πρότυπα που να εξασφαλίσουμε τη σωστή διαδικασία Έχουμε 27 διαδικασίες χωριστές, διαφορετικές για την ε, ανακύκλωση στην Ευρώπη, γιατί οι τεχνοκράτες και οι πανεπιστημιακοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα θέματα αυτά. Η Αυστρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης και μια θαυμάσια νότια χώρα της Ευρώπης έχει το χαμηλότερο ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Μια άλλη παλιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια αντιμετώπιση η οποία είναι τελείως διαφορετική σε ποσοτικό επίπεδο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να γίνεται κάποια προσπάθεια για να θεσπιστούν κοινοί ε, κανόνες και κοινέ προδιαγραφές. Εσείς και οι τρεις μιλήσατε για τις παράνομες εξαγωγές. Αλλά είναι ο καιρός να σκεφτούμε ότι για πάρα πολλούς τα ηλεκτρονικά στοιχεία των υπολογιστών θεωρούνται από πολλού ω απλώ απόβλητα. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίηση πολλών αυτών. Έχουμε πάρα πολλά κοντέινερ τα οποία εξάγουν προϊόντα τα οποία είναι ε, παράνομα από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν οι εξαγωγείς ότι απαγορεύεται η εξαγωγή αυτών των υλών οι οποίες είναι αναχρησιμοποιήσιμες. Πιστεύω ότι έχουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο το οποίο θα αποτρέψει την, θα αποτρέψει την ε, εξαγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, αλλά πρέπει να κλείσουμε και τα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό είναι εξάλλου πολύ σημαντική και μας ενδιαφέρει επίσης και η χρήση πρώτων υλών από, του, το, από τους στρατιωτικούς και, και εκεί πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση των πραγμάτων. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν μας έχει παρουσιάσει ακόμα τις προτάσεις και δεν είναι παρούσα να μας πει κάτι για την πολιτική βιομηχανία. Θα πρέπει να κάνουμε σαφές στην Κομισιόν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι προοπτικές από την πλευρά αυτή της Επιτροπής αν μπορούμε λοιπόν μαζί με τον κύριο πίτροπο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα, κάτι το οποίο φαίνεται να δυσκολεύει την Κομισιόν, θα προχωρήσουμε σε μια αποτελεσματική βιομηχανική και πολιτική περιβάλλοντος. Ο κύριος Λάμπερτ. Να συνεχίσω από όσα υπόθηκαν. Κύριε Σώμα, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει νομοθεσία, αλλά λείπει η εφαρμογή της. Συμφωνούν όλοι οι ομιλητές από αυτού ή υπάρχουν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να πληρώσουμε στην νομοθεσία μας, όπως ε, είπε ο προηγούμενος άδερφος, ο κ. Φλόρενς. Φαίνεται να οδεύουμε αργά προς κανόνες ε, και νομοθεσία για ενεργειακή απόδοση. Και πάλι απευθύνομαι και στους τρεις ομιλητές. Θεωρεί κανείς από εσά ότι πρέπει να έχουμε κανόνες και στόχους για αποδοστικότητα πόρων ή είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Προς τον κύριο Αρντίτη, μου άρεσε το γεγονός ότι επιστήσατε την προσοχή στη ζήτηση και όχι μόνο στην ε, ε, προμήθεια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και τα ε, το πώς λειτουργεί η ζήτηση. Τι προτάσεις έχετε να κάνετε για την ε, νομοθετική μας δράση. Θα πρέπει να το κάνουμε μέσω φορολογίας, μέσω μηχανισμών που θα βασίζονται στην αγορά. Έχετε κάποιες προτάσεις να μας κάνετε. Και τρίτον προς τον κύριο Μάγερ, Είδαμε τι ε, αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου για τη χρήση των γεών και τι λύσεις ε, θεωρείτε ότι ε, υπάρχουν επ' αυτού και αν υπάρχει κάποιο εφεδρικό σχέδιο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ο κύριος Τσιμάνσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να διορθώσω κάτι, καταρχάς. Δεν είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσβαση σε πόρους. Έχουμε από τις μεγαλύτερες ε, ε, αποθέματα αργύρου και χαλκού παγκοσμίου. Και όταν εξάγουμε άργυρο μπορούμε να εξάγουμε και άλλους πόρους, ε, όπως και σπάνιες γέες. Κάνω έκκληση λοιπόν προς όλους μας να εκτιμήσουμε αυτά τα οποία έχουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκε μία λανθασμένη εναλλακτική λύση ε, για την ανακύκλωση και το διεθνές εμπόριο ιδιών πόρων. Δεν είναι αλήθεια ότι πρέπει να επιλέξουμε έναν πυλώνα ε, και να ακολουθήσουμε μία άγουσα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τους τρεις πυλώνες. Και το να ζητούμε τη μείωση της κατανάλωσης είναι μη ρεαλιστικό, αλλά είναι και επικίνδυνο. Διότι αυτό σημαίνει ότι θα μειώσουμε τη βιομηχανική μας δραστηριότητα. Επίσης σημαίνει ότι θα ε, περιορίσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε και διαρροή εγκεφάλων στη συνέχεια και ε, αυτοί που ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη θα αρχίσουν να αναζητούν ε, τη γη της επαγγελίας αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο προσεκτικοί για... όταν ζητάτε μείωση της κατανάλωσης και καλύτερη διαχείριση. Thank you, Chair. Η κυρία Μέρκη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους. Συμφωνώ κύριε Αρντίτη ότι εστιάζεται την προσοχή σας στην κατανάλωση και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας ως προς την κατανάλωση. Ορισμένες φορές φοβούμε ότι ασχολούμαστε πολύ με την νομοθεσία και δεν δίνουμε κίνητρα, διότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι από το να ε, υποχρεώνουμε κάποιους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Ίσως θα μπορούσαν να έχουμε κατάλληλα ερεθίσματα για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε. Επίσης, μου αρέσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι επικεντρωθήκατε στην επαναχρησιμοποίηση, διότι ορισμένες φορές έχουμε μια τάση να πετάμε τα πάντα στα σκουπίδια και να ξεκινούμε ε, με καινούρια πράγματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος και πώς το ε, βλέπετε εσείς ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Επαναχρησιμοποίηση των υλικών με την έννοια ότι ναι μεν κατανοητό ότι μπορεί να θέλουμε να έχουμε κάτι που να είναι ενεργειακά αποδοτικό ή καλύτερο για το περιβάλλον μας, αλλά ίσως θα μπορούσε να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην ε, κατασκευάζεται μια συσκευή εκ του μηδενός, αλλά να πάρετε μια παλιά συσκευή και να τη βελτιώσετε σε κάτι που θα είναι πιο καλέσθητο, καλύτερο, πιο γρήγορο. Ε, και να υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση στην ανακύκλωση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που με ανησυχούν. Ε, μιλάμε πάντα για τα ίδια υλικά και για μένα υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξίας ε, της χρήσης ενός iPhone αν θέλετε και ενός ανεμόμυλου. Ξέρουμε ότι όλοι θέλουμε να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, αλλά αν ένας ανεμόμυλος χρησιμοποιεί τις ίδιες ύλε που έχουμε και σε ένα iPhone, τότε εγώ θα μείωνα τον ανεμόμυλο. Αλλά επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να έχουν ένα iPhone, τι θα γίνει με τον αγώνα για τις ίδιες ύλε. Ποιος θα καθορίζει λίγο πολύ ποιο θα παίρνει τι, η αγορά θα το καθορίζει. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει και μια κάποια ε, ταξινόμηση. Ποια είναι η καλύτερη χρήση ε, η πιο πολύτιμη χρήση για ένα υλικό. Δεν λέω ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε την ταξινόμηση, αλλά όταν μιλάμε για παράδειγμα για άλλους πόρους, όχι για τις σπάνιες γεές για παράδειγμα, αλλά για τη βιομάζα, όλοι θέλουν ε, βιομάζα, θέλουν για την ενέργεια, για τη φαρμακευτική, για βιοδιασπόμενα προϊόντα. Ποιος λοιπόν θα την πάρει τη βιομάζα. Για μένα λοιπόν το ερώτημα είναι πώς θα ε, στήσουμε ένα σύστημα όπου ο καθένας θα λαμβάνει αυτό που θέλει και δεν θα γίνεται αγώνας για να λάβουμε όλα τα ίδια προϊόντα. Για να ξανάρθω τώρα στο θέμα της ανακύκλωσης. Αν η Ευρώπη εξαρτάται τόσο πολύ από τις εξαγωγές, αλλά εξάγει τόσο πολλά παλιοσίδερα, ε, ξέρω ότι δεν μπορούμε να στραφούμε ενάντια στους κανόνες του ΠΟΕ, αλλά μήπως υπάρχει τρόπος να προλάβουμε τις εξαγωγές δίνοντας νέα όθηση στην ευθύνη των παραγωγών, απαιτώντα λοιπόν μέσω νομοθεσίες ε, από τους παραγωγούς να αποσύρουν οτιδήποτε διαθέτουν στην αγορά. Έτσι θα κλείσει η πόρτα για τις εξαγωγές στην Ευρώπη, θα ανακυκλώνονται τα πάντα και θα έχουμε ε, μια κοινωνία όπως αυτή που επιθυμούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις. Νομίζω φτάνουν οι ερωτήσεις τώρα για να μπορέσουμε να ε, έχουμε τις απαντήσεις και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. κύριος Τσόμα, το λέω σωστά το όνομά σας, Τσόμα, μάλιστα. Ευχαριστώ. για την ερώτησή σας ε, για την ανακύκλωση, αν είναι βιώσιμη οικονομικά σήμερα και το παράδειγμα του λιθίου και τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πιθανή οδοί. Έχουμε δουλέψει με τη Eurometal, την Ευρωπαϊκή Ένωση Μετάλλων, ε, για κάποιες προτάσεις για το θέμα των πρώτων υλών και η πρόταση που προκύπτει από αυτή τη δουλειά μας με τη Eurometal και από το Ινστιτούτο με το οποίο συνεργαστήκαμε είναι ότι καταρχήν χρειάζεται έρευνα για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι οικονομικά ανακυκλώσιμα για να βελτιώσουμε την τεχνολογία σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Δεύτερον, μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από το σύστημα ανάκτησης των προϊόντων και είπα και στην παρέμβασή μου ότι κάνουμε ανακύκλωση λαμβάνοντας υπόψη και τον όγκο και την αξία των υλικών και τα επικίνδυνα υλικά. Έχουμε οργανώσει σύστημα ε, για την ε, παράδοση των υλικών μετά τη χρήση τους, ε, ώστε να έχουμε ανάκτηση των επικίνδυνων υλικών, αλλά για τα επικίνδυνα υλικά θα μπορούσε να επεκταθεί το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται και να συμπεριλάβει και άλλα κρίσιμα υλικά που σήμερα δεν είναι από οικονομικής πλευράς ανακυκλώσιμα. Για τον οικολογικό σχεδιασμό θα επανέλθω σε κάτι που ανέφερα προηγουμένως, ε, είπα ότι έχουμε ένα κύκλο στην οικονομία. Η βιομηχανία Μα μας ε, βρίσκεται και στην αρχή και στο τέλος της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Εμείς παρέχουμε τα υλικά. Εγώ μίλησα για την ανακύκλωση και για τον τρίτο πυλώνα της πρωτοβουλίας ε, για τις πρώτες και οι άλλοι δύο πυλώνες είναι εξίσου σημαντικοί, αν και εγώ δεν ε, εστιάστηκα στην παρέμβασή μου σε αυτούς τους άλλους πυλώνες. Η βιομηχανία μας ε, προμηθεύει τα υλικά που μπαίνουν ε, τα προϊόντα των κατασκευαστών άμεσα ή έμεσα, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα ή άλλο είδος εξοπλισμό και προσπαθούμε να πάρουμε τα προϊόντα τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους και να τα ανακυκλώσουμε για να ανακτήσουμε τα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα προϊόντα και να τα μεταποιήσουμε σε νέα προϊόντα ή υλικά τα οποία και πάλι θα χρησιμοποιήσουν στον εξοπλισμό τους. Για να το κάνουμε αυτό, είναι σαφές ότι όσο περισσότερο δουλέψουμε πάνω στην ανακύκλωση στην, μέσα στο πλαίσιο της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, τόσο περισσότερο θα συμμετέχουμε στην ανάπτυξη προϊόντων. Και τόσο πιο εύκολο θα είναι να τα ανακυκλώσουμε. Το iPad, παραδείγματος στην αρχή δεν μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την μπαταρία από το iPad, αλλά στην ανακύκλωση πρέπει να μπορείς να βγάλεις την μπαταρία. Ήταν κάτι πολύ απλό που δεν το είχαν σκεφτεί η παραγωγή του iPad. Ένα από τα βασικά λοιπόν σημεία είναι να συμμετέχουμε στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για να εξασφαλίσουμε σωστή ανακύκλωση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για τις παράνομες εξαγωγές τι λύσεις υπάρχουν. Καταρχήν πιστεύουμε ότι μπορεί ο τελωνιακός κώδικας ε, να βελτιωθεί, να προσθέσουμε πληροφορίες στις τελωνιακές ε, διασαφήσεις για να μπορέσουν οι τελωνιακοί να καταλάβουν τι είναι πρωτογενές τι, αποτελεί επανάχρηση και τι είναι πρωτότυπο, πρωτότυπος εξοπλισμός. Γιατί πολύ συχνά η επανάχρηση χρησιμοποιείται ως ψευδής δήλωση η βασική πρόταση που κάναμε με τη Eurometal είναι μια πιστοποίηση ε, της τελικής μονάδας ανακύκλωσης, όπου και αν βρίσκεται, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού. Αυτή η πιστοποίηση της μονάδας ανακύκλωσης θα καλύπτει και περιβαλλοντικά στοιχεία και στοιχεία υγείας και ασφάλειας ε, και λειτουργικά κριτήρια. Δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκο, πρέπει να διασφαλίζει τα ελάχιστα κριτήρια ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η ανακύκλωση και με σωστούς περιβαλλοντικούς όρους και διασφαλίζοντας τη μέγιστη ανάκτηση υλικών. Από τη συζήτηση που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους διαμορφώνοντες στην πολιτική, αυτή η πρόταση δεν φαίνεται να είναι παράλογη. Υπάρχουν οι κανόνες του ΠΟΕ, αλλά είναι υπομελέτη αυτή η πρόταση. Πιστεύουμε ότι θα είναι τεράστια η αλλαγή, γιατί η εξαγωγής των παλιοσίδερων θα είναι υπεύθυνη και για την τελική ανακύκλωση των προϊόντων. Για την ερώτηση του κυρίου Λαμπέρτ σχετικά με τα κενά που υπάρχουν, σαφώ υπάρχουν κενά και ίσω δεν τα παρουσίασα εγώ επαρκώ στην παρέμβασή μου. Πιστεύουμε ότι αν η υφιστάμενη νομοθεσία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σωστά, θα είχαμε ήδη βελτιώσει δραματικά την ε, ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση στην Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κενά, ιδίω στου στόχους που έχουμε για τη συλλογή. Αν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη συλλογή των ε, υλικών, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και, ε, όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα των ε, υλικών που συλλέγουμε. Έγινε μια ερώτηση για την έρευνα και ανάπτυξη και τον κίνδυνο του να μειώσουμε την ε, έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Συμφωνώ με την άποψή σας και πιστεύω ότι η ανακύκλωση προσφέρει τεράστιο δυναμικό για να αναπτύξουμε περαιτέρω τη βιομηχανία στην Ευρώπη με νέες επενδύσεις και με θέσεις απασχόλησης, όχι μόνο για ε, αυτούς που θα δουλεύουν στις βιομηχανίες αυτές, αλλά και για την έρευνα και ανάπτυξη που θα είναι απαραίτητη για αυτόν τον τομέα. Και για την ε, αναχρησιμοποίηση πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η προτιμόμενη λύση. Θέλουμε ε, τελικά να έχουμε επαναχρησιμοποίηση του υλικού που περιέχεται στο προϊόν, όχι να χάνεται το περιεχόμενο αν δεν χρησιμοποιείται εκ νέου το προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής, της, ζωής του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαρντιτή, σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να οργανώσω καλύτερα την απάντησή μου σε δύο τμήματα. Πρώτα το θέμα της κατανάλωσης. Πρέπει να διαλύσω μια παρεξήγηση. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να μην χρησιμοποιήσουμε τον τρίτο πυλώνα. Αλλά λέω ότι αν δώσουμε προτεραιότητα στον τρίτο πυλώνα, στην κατανάλωση των πόρων, και τον τρόπο αντιμετώπισης των αποβλήτων, μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για τον πρώτο και για τον δεύτερο πυλώνα. Είναι πολύ διαφορετικό από το να πούμε ότι δεν το χρειαζόμαστε τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Απλώς θα πρέπει να τους χρησιμοποιούμε εκεί που τις χρειαζόμαστε. Για την κατανάλωση των πρώτων υλών θέλω επίσης να διαλύσω άλλη μια παρεξήγηση. Δεν λέω μονάχα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πτυχή των, των προβλημάτων είπα ότι πρέπει η βιομηχανία να αντιμετωπίσει την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων και την οικολογική αποδοτικότητα. Όλα αυτά οδήγησαν σε σημαντική καινοτομία και καλύτερη χρήση από τη βιομηχανία. Η μείωση λοιπόν της κατανάλωσης των πόρων δεν μιλάμε για τον τελικό καταναλωτή μονάχα, μιλάμε για την οικολογική αποδοτικότητα στις βιομηχανίες. Αυτό μας δίνει ένα τεράστιο δυναμικό δράσης σε επίπεδο έρευνα και ανάπτυξη και σε επίπεδο βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να παραμελήσουμε όμως και το, τα σχήματα κατανάλωση. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να νομοθετούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξει ο τρόπος κατανάλωσης και τα σχήματα κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά η νομοθεσία μπορεί να επηρεάσει αυτά τα σχήματα κατανάλωσης. Και είναι σημαντική αυτή η διάσταση της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων. Παραδείγματος χάρη στην επαναδιαμόρφωση της οδηγίας για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να θεσπίσουμε συγκεκριμένους στόχους επαναχρησιμοποίησης. Σε κάποια κρατημέλη αυτό μπορεί να ήταν δύσκολο στην πράξη, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα παράδειγμα μέσα από το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο κατανάλωσης. <clears throat> Και από την οικολογική σχεδίαση, εμείς τώρα αντιμετωπίζουμε πολλά προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα παρόμοια με υπολογιστέ. Ε, όχι μόνο υπολογιστέ, αλλά εκτυπωτέ, ε, παιχνίδια ηλεκτρονικά. Όλα αυτά περιλαμβάνουν σπάνιες γιές και σπάνια μέταλλα τα οποία πρέπει να ανακτηθούν. Αλλά το ερώτημά μου είναι τι μπορούμε να πούμε ως προϋπόθεση για την παραγωγή αυτών των προϊόντων από πτυχή πόρων. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή απολύτως τίποτα, τίποτα δεν έχει γίνει. Και πάλι λοιπόν μπορούμε να δούμε να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τόσο το σχήμα κατανάλωσης για στόχους ε, ανάκτησης και την αποδοτικότητα χρησιμοποίησης στη βιομηχανία μέσω της οικολογικής σχεδίασης. Όλα αυτά με οδηγούν στο δεύτερο ερώτημα. για τα χάσματα τα οποία, τα κενά τα οποία υπάρχουν στην νομοθεσία και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Το παράδειγμα της οικολογικής σχεδίασης είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, όπου είναι φανερό ότι χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες είναι στη διάθεσή μας. Μια άλλη οδηγία που θα ψηφίσετε στις 3 Φεβρουαρίου είναι η οδηγία WE, και εκεί πάλι πρέπει να δώσουμε σημασία στο να έχουμε στόχους συλλογής οι οποίοι είναι φιλόδοξοι. <clears throat> Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, αυτό υπονομεύει τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται για την ανακύκλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και κάποιες καινοτόμες πρακτικές οι οποίες προτείνονται από τις οδηγίες αυτές. Αυτό με οδηγεί να αντιμετωπίσουμε και τα μη νομοθετικά εργαλεία ή τουλάχιστον τα ήπια νομοθετικά εργαλεία και τις προτροπές προς την αγορά. Στην οδηγία αυτή προτείναμε να ενισχυθεί η λεγόμενη ευθύνη του μεμονωμένου παραγωγού. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους κατασκευαστές να παράγουν προϊόντα τα οποία είναι πιο εύκολα αποδομήσιμα. Και εδώ πάλι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να καινοτομήσουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθεί στην νομοθεσία ένα εργαλείο για την αγορά. Και αν μιλάμε για την οικολογική σχεδίαση, είναι πάλι μια παρόμοια κατάσταση. Γιατί ξέρουμε ότι το να χρησιμοποιήσουμε ανακυκλωμένα υλικά εξοικονομεί πολλέ εκπομπές διοξιδίου του άνθρακο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αμοιβών και κυρώσεων, λέγοντα ότι έχετε αυτές τις προδιαγραφές για ενεργειακή αποδοτικότητα. Αν χρησιμοποιείτε όμως την ανακύκλωση σε κάποιο βαθμό, εμείς εκτιμούμε ότι μειώνεται και τη συνολική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος από το προϊόν αυτό σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Επομένως μπορούμε να σας ανταμείψουμε σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Ένας τρόπος ακόμα λοιπόν να καιροτομήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την νομοθεσία που αφορά τις απαιτήσει του περιβάλλοντος και μια ανταμοιβή σε επίπεδο αγοράς. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε ρυθμίσεις πανευρωπαϊκές για το θέμα αυτό είναι το θέμα της φορολογίας των πόρων αυτών, των πρώτων υλών ή αν δεν σας αρέσει η έννοια της ε, φορολογίας, το πώς μπορούμε να καταβάλουμε το αντίτιμο για την απόκτηση των πρώτων υλών. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα της εργασίας υπήρξε, ήταν πολύ ψηλή τα τελευταία 30 χρόνια γιατί υπήρχε και μια σωστή φορολόγηση του συντελεστή εργασίας. Γιατί να μην σκεφτούμε και ένα αντίστοιχο σύστημα για, τους πρώτου, για τις πρώτες ύλε και ίσως αυτό θα ενισχύσει ιδιαίτερα την αποδοτικότητα των πρώτων υλών, της χρήσης των πρώτων υλών ετέθηκε το ερώτημα αν μπορούμε να θεσπίσουμε στόχους, όπως έχουμε στόχους για αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας, να έχουμε στόχους για την αποδοτικότητα των ε, πρώτων υλών. Ξέρετε ότι εμείς υποστηρίζουμε να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για την χρήση ενέργειας και των πρώτων υλών, γιατί μόνο οι δεσμευτικοί στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να γίνουν σωστές προϋποθέσεις σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αυτό όμως δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, γιατί αν έχετε <clears throat> νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ανάγκη να υπάρχουν εξοικονομήσεις στους, στις πρώτες θα γίνει αυτό από τη βιομηχανία. Αν πείτε ότι α, καλό είναι αυτό να κάνουμε εξοικονομήσεις και να έχουμε απόδοση, πώς μπορεί η βιομηχανία να εξασφαλίσει ότι θα έχει τη σωστή απόδοση σε παιδί τους. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η, η όθηση σε νομικό επίπεδο. Και αυτό μπορεί να γίνει για, τις πρώτους, για τις πρώτες ύλες. Αλλά αν το κάνουμε αυτό για τις πρώτες ύλες, όπως έλεγε και μια διαφάνεια δικιά μου, θα πρέπει να δούμε το συνολικό αντίκτυπο στην κατανάλωση πρώτων υλών, που περιλαμβάνει τον αντίκτυπο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά το λεγόμενο σακίδιο του περιβάλλοντος, δηλαδή την, τον αντίκτυπο σε υλικά τα οποία μένουν αχρησιμοποιητά. Και εδώ η εξόριξη είναι κάτι το πολύ καλό παράδειγμα. Όταν εξορίσουμε για να βγάλουμε κάποιο χρήσιμο υλικό, δημιουργούμε και πάρα πολλά εξορυκτικά απόβλητα, που είναι περίπου 20 με 25% από τα συνολικά μας απόβλητα, που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Δεν επαναχρησιμοποιούνται τουλάχιστον. Οι στόχοι λοιπόν <clears throat> για την ε, αποδοτικότητα των πρώτων υλών, δεσμευτικοί αλλά που να συνδέονται με, το συνολικό, με τις συνολικές απαιτήσει για το υλικό το οποίο πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Μάιρ, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα. Το REACH για την ε, βιομηχανία. Εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια αξιολόγηση για το πόσο μας επηρεάζει. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα αυτό και σε κάποιο βαθμό έχει περιπλέξει τη χρήση πρώτων υλών και έχει μειώσει κάπως την ασφάλεια εφοδιασμού για την εμπορική πολιτική βεβαίως. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις διμερείς συμφωνίες στον εμπορικό τομέα να μιλήσουμε και για περιορισμούς εξαγωγών, το κάναμε αυτό με την ε, Ουκρανία, είπαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί εξαγωγών, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε και μέσα, όπως ελέγχθη, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και να πούμε ότι αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, τότε θα πρέπει να μην έχετε περιορισμούς εξαγωγών πρώτων υλών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. για την ανακύκλωση και την παρεμπόδιση των παρανομών εξαγωγών. Εγώ πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή των κριτηρίων και των κανόνων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα είναι η οδηγία για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θεσπίζονται. Και εδώ το άχθος της απόδειξης θα πρέπει να βρίσκεται στους εξαγωγείς. Αυτοί θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι σωστή η εξαγωγή αυτών των προϊόντων και θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Τα κρίσιμα και στρατηγικά υλικά, οι πρώτες ύλε μάλλον. Κανένα από τα στρατηγικά υλικά που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στην Γερμανία ή στην Ευρώπη και τα στρατηγικά υλικά. Το κριτήριο για αυτά τα υλικά θα πρέπει να είναι και η υπερσυγκέντρωσή τους σε ορισμένες χώρες που είναι από πολιτική άποψη εύθραυστες χώρες. Αναφέρθηκε το θέμα του ότι μπορούμε να ανακτήσουμε πάρα πολλά, να αποκτήσουμε πάρα πολλά σπάνια υλικά από την εξόριξη ε, χαλκού και αργύρου. Και ξέρω ότι έμαθα μάλιστα ότι στην περιοχή του Φλένσπορκ στην Βόρεια Γερμανία υπάρχουν και σημαντικά κοιτάσματα ε, σπανίων γεών. Ίσως με μελλοντικές ε, τεχνολογίες μπορούμε κάτι, ένα υλικό το οποίο δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ως στρατηγικού χαρακτήρα να αποκτήσει αυτό το χαρακτηρισμό στο μέλλον. Βέβαια η, βιομηχανία στη Γερμανία ανησυχεί τα μάλα με τον περιορισμό εξαγωγών σπανίων γεών από, ε, από την Κίνα για τις σπάνιες γεές. Αν υπάρχει τώρα εναλλακτικό σχέδιο, υπάρχουν πολλές ε, σκέψεις στην ε, Γερμανία να σκεφτούμε άλλες πηγές που δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν υπάρχει μια προσπάθεια από τη γερμανική κυβέρνηση να υπάρξει μια καλύτερη διαφοροποίηση για την ε, πρόσβαση σε, πράσ... σε σπάσινες γέες με το να δημιουργηθούν νέες εμπορικές σχέσεις με άλλους φορείς, παραδείγματος χάρη η Μογγολία, το Καζακστάν είναι χώρες με τις οποίες πρέπει να διαρευνηθούν οι δυνατότητες εμπορικών συμφωνιών για αυτές τις ε, πρώτες ύλες και επομένως υπάρχουν τέτοιου είδους δυνατότητες διαφοροποίησης. Δεύτερος γύρος τώρα. Κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομα ερωτήματα κατανόησης για να καταλάβουμε και από πολιτικής πλευράς πώς πρέπει να το χειριστούμε. Όσον αφορά τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων ε, ηλεκτρικών και παλιοθυδερών, καταρχήν υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε για την μαύρη αγορά να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα, είναι μεσαία σοβαρότητα στο πρόβλημα, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει δυνατότητα οι τελωνιακοί να ελέγχουν πιο εύκολα τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο μέσω της τελωνιακής διασάφησης. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ε, ή όχι και υπάρχουν ε, ε, ενδεχομένως προτάσεις για την αντιμετώπιση, την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Ποια είναι η αιτία για την οποία υπάρχει αυτό το παράνομο εμπόριο τέτοιων υλών από την Ευρώπη. Ακόμη θα ήθελα να ρωτήσω για τις ε, πρώτες ύλες ε, από την, ε, που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τα εμπόδια στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες Ποια είναι, είναι διοικητικά εμπόδια, κάποιες χώρες θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες, υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρεζίνα. Ευχαριστώ. Ε, άκουσα αυτά που είπατε για την ανακύκλωση και συμφωνώ και εγώ προσωπικά για αυτά που είπατε για την ανακύκλωση. Πιστεύω ότι η ανακύκλωση είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι και να είμαστε και πρωτοπόροι σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη πιστεύω ότι όταν κάνουμε μια συζήτηση για τις πρώτες ύλε. αυτό είναι ένα θέμα που είναι παράπλευρο σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που έχει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η ανακύκλωση αποτελεί ευκαιρία για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία. Νομίζω ότι το πρόβλημα προκύπτει όταν μιλάμε για πρώτες ύλες, νέα μέταλλα, νέες πρώτες ύλες ε, που δεν βρίσκουμε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να τις προμηθευτούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν με πολιτικά μέσα και πρέπει να ζητήσουμε ίση πρόσβαση στις αγορές ε, τρίτων χωρών. Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν είναι η μόνη χώρα που έχει να λύσει τέτοιο πρόβλημα σε σχέση με τις πρώτες ύλε. Αν δούμε και τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπάθησαν να το λύσουν αυτό το πρόβλημα με, το ότι ε, συγκεντρώνουν πρώτες ύλε και τις ισορεύουν μέσα στη χώρα τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να έχουν αποθηκευμένες πρώτες ύλε οι οποίες μελλοντικά θα χρειαστούν. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, Stockpiling Act, θα μπορούσαμε και στην Ευρώπη να έχουμε μια αντίστοιχη στρατηγική και να μην έχουμε 27 διαφορετικές στρατηγικές για τις πρώτες ύλες. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αγορά των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόμοιο με αυτό το οποίο κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, με την ομοθεσία τους ε, για τη δημιουργία αποθεμάτων ε, πρώτων υλών. Διαφορετικά θα διατρέχουμε τον κίνδυνο των μέτρων που θα λαμβάνουν χώρες όπως η Κίνα ή η Αφρική ή η Ινδία. δεν μπορούμε ο καθένας μόνος του να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ευγενών μετάλλων και των σπανίων γεών. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο και η Κίνα έχει συμβάλει μέσω εμποδίων στις εξαγωγές της. αλλά και εμείς ως Δύση και ως δυτικός πολιτισμός έχουμε συμβάλει στη δημιουργία του προβλήματος γιατί μερικές φορές ε, ε, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην προστασία της φύσης από ότι στη στρατηγική εξασφάλιση τέτοιων πρώτων υλών. Υπάρχουν χώροι και στην Ευρώπη στην οποία ε, υπάρχουν ε, ευγενή μέταλλα και στην, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει την κρίση από μόνοι μας και μπορούμε να δούμε τις λύσεις που έχουν βρει οι Αμερικανοί γιατί και στις ΗΠΑ και στο Βιετνάμ έχουν δημιουργηθεί τέτοιοι χώροι αποθήκευσης. Και να μην δημιουργούμε ένα μύθο σχετικά με τα ευγενή μέταλλα, αν υπάρχουν λύσεις δεν ε, περιορίζονται οι δυνατότητές μας μόνο στις εισαγωγές από την Κίνα. Πρέπει να δούμε και κατά πόσο έχουμε εμείς δημιουργήσει το πρόβλημα. θα βρίσκεται μονίμως σε κρίση η βιομηχανία μας αν δεν λάβουμε δραστικά μέτρα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για την ε, σαφέστατη περιγραφή για το πέρασμα από το waste business το high-tech business το θέμα της ανακύκλωσης και νομίζω ότι δόθηκαν και εξαιρετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις ε, οι οποίες έγιναν εδώ από τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να σας πω ότι πράγματι πρέπει να γίνει ένα συνδυασμός όλων αυτών με βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη. Είναι εξαιρετικά τα όλα όσα γίνονται. Ακούσαμε ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες συγκεκριμένε προτεραιότητες, θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς όταν αναφερόμαστε σε πρώτες ύλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Αλλά αν εσείς μπορούσατε να καθορίσετε τις πρώτες ύλε σε αυτό το πλαίσιο, ώστε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ επικεντρωμένοι Τι θα λέγατε, πώς θα προχωρούσατε το θέμα αυτό. Κυρία Μέρκης. Van ε, ε, schaarse materialen. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ε, τι γίνεται με τις ε, σπάνιες γεές και τα σπάνια υλικά. Το συζητήσαμε μεν, αλλά όταν μιλάμε για πρώτες ύλε δεν αναφερόμαστε μόνο στις σπάνιες γεές, αναφερόμαστε και στη βιομάζα Ε, και σε άλλα ε, υλικά τα οποία είναι περιζήτητα. Όσον αφορά τα ορυκτά, νομίζω ότι επικεντρωθήκαμε μόνο στα σπάνια. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στο εξής. Θέλουμε να έχουμε πρώτες ύλες και σπάνια σε κάποια περίπτωση. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν πιο χρήσιμο να τα χρησιμοποιούμε με άλλο τρόπο και αυτό φυσικά ε, μας οδηγεί σε γνωστά προβλήματα. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα καθαρό κινητήρα, ίσως γιατί αυτό δεν είναι ενδιαφέρον για το καταναλωτή. Ή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αιωλικό πάρκο, διότι το ίδιο υλικό που χρειάζεται για την κατασκευή του χρησιμοποιείται σε άλλα προϊόντα που ε, ενδιαφέρουν περισσότερους καταναλωτές. Τα ακούσαμε αυτό. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να νομοθετήσουμε ή τουλάχιστον να κάνουμε μια κατάλληλη ταξινόμηση για τη χρήση αυτών των σπανιότερων υλικών. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Φαμπρέντ. Ζητώ συγγνώμη, ε, δεν άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά το θέμα της οδηγίας ε, Wii για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Αναφέρθηκε τι θα μπορούσαν να κάνουν οι αρχές αλλά και ο κλάδος επί του θέματος. Αυτό το έχουμε συζητήσει, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια ψηφοφορία ε, που βρίσκει σύμφωνο σχεδόν όλο το κοινοβούλιο. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια επί του θέματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ε, ψηφίσουμε σωστά την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φιλόδοξοι στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτή την οδηγία και μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να περιορίσουμε κατά πολύ τις εξαγωγές. Επομένως θα μπορέσουμε ίσως να αποφύγουμε ε, την ε, μαζική απόρριψη των αποβλήτων αυτών σε τρίτες χώρες. Ε, το πρόβλημα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις μέρες μας είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την απόρριψη αυτής της νομοθετικής πράξης. Κύριε Σώμα, ζητώ συγγνώμη αν προφέρω και λάθος το όνομά σας. Γνωρίζω ότι ε, εκπροσωπείται τη Unicorn, μια ε, επιχείρηση την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Συχνά υπάρχουν ε, πολλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στις ε, χώρες μέλη υπάρχουν μεγάλες πιέσεις και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. ένα αποτελεσματικό εφεδρικό σχέδιο, δηλαδή επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ. θα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και η νομοθετική στήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε δύο λεπτά σε κάθε ομιλητή χρόνο να απαντήσει σε αυτό το γύρο των απαντήσεων. Κύριε Τσόμα, ξεκινήστε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. για το θέμα των δεδομένων για τις παράνομες εξαγωγές. Επειδή είναι παράνομες, προφανώς δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Θα σας παραπέμψω στην Ίμπελ. Η Ίμπελ έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά επί του θέματος και μας έχει δώσει πολύτιμες πληροφορίες μέσω διαφόρων δοκιμών που έχουν κάνει ε, και ε, βρήκαν στα σύνορά μας ε, τεράστιες ποσότητες παρανομιλικού που εξάγεται στα μέσω και βοηθείων. Ένας άλλος τρόπος να το αξιολογήσουμε, κάτι το οποίο είναι και λίγο πιο ε, επαφές, είναι να επισκεφτούμε τους λιμένες που λαμβάνουν τα υλικά ε, και να δούμε κατά πόσον το ανακυκλούμενο υλικό είναι όντως ανακυκλούμενο για να δούμε τι ακριβώς εξάγεται. Εμείς εκτιμούμε ότι ε, είναι πάνω από το 40% το ποσοστό. Βέβαια πρόκειται για εκτίμηση, αλλά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ε, σαφώς θα πρέπει οι τελωνιακές αρχές να επικεντρώνονται και στο τι, εξάγεται, ε, τι εισάγεται αλλά και το στο τι εξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικές πολιτικές ε, για τα υλικά αυτά. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω εντάχει ε, το θέμα των σπάνιων γεών. Ίσως εμείς να δημιουργήσαμε πρόβλημα με τις σπάνιες γεές, ε, ως εμείς εννοώ τις χώρες εκτός της Κίνας που έχουν ε, αποθέματα σπάνιων γεών, ε, και αυτή τη στιγμή η Κίνα χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα με εμά για να μειώσουν τις εξαγωγές και λένε ότι θέλουν να βελτιώσουν τα ορυχεία τους. Είναι θέμα ισότιμου πεδίου και το ίδιο ισχύει και ε, με τους στόχους που θέλουμε να θέσουμε. Το γεγονός ότι έχουμε, θέλουμε να έχουμε ένα υποχρεωτικό πλαίσιο είναι να αποφύγουμε να ξανασυμβεί το ίδιο. Ε, διότι θα φτάσει μια στιγμή που όλα τα υλικά θα πηγαίνουν σε μη ε, υγιή, μη μη φιλικά ως προς το περιβάλλον ε, μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουν το ίδιο ε, πρόβλημα. Επομένως, είτε μιλάμε για πρώτες είτε για δευτερεύουσες ύλε, το να υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το γουί, νομίζω ότι θα σταματήσω τώρα ως προς το να πείσουμε τα κράτη-μέλη, κυρίως για την εφαρμογή της νομοθεσίας στα σύνορα και στους λιμένες, ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει ε, να προσδώσουν το αντίστοιχο βάρος σε αυτή τη διαδικασία. Και συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαρντιτή, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι η ασφάλεια των, του εφοδιασμού για σπάνιους πόρους ισχύει εδώ και πολύ καιρό και είναι μια μακροχρόνια προοπτική. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η δυσκολία πρόσβαση σε σπάνια, σπάνιες πρώτες και η βιομάζα στο τέλος θα γίνει και αυτή ένας κρίσιμος και σπάνιος πόρος. Τονίζω για αυτό τον λόγο ότι πρέπει να υπάρξει καινοτομία από τις επιχειρήσεις σε το, στο μοντέλο του επιχειρήν και στο μοντέλο της ανάπτυξης. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι σπάνιες γης, αύριο όμως θα είναι βιομάζα και άλλοι πόροι. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξουν μια σωστή ισορροπία μεταξύ απόκτησης πρώτων υλών και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σωστό αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορούμε να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο αναγκών. Η Κομισιόν έχει αρχίσει να απαντάει το θέμα αυτό λέγοντας ότι έχουμε εδώ ένα κατάλογο κρισίμων πρώτων υλών και κανένα υλικό σε αυτά το κατάλογο δεν μπορεί να βρεθεί με τόση ευκολία στην Ευρώπη με άλλο τρόπο παρά μόνο με την ανακύκλωση των αποβλήτων. Επομένως, αυτό χρειάζεται στην Ευρώπη σήμερα, να, να χρησιμοποιήσουμε τα αστικά απόβλητα για ανακύκλωση. Σήμερα λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση. Εκεί υπάρχει πραγματικό δυναμικό και δυνατότητα ανάκτησης των ε, σπανίων αυτών πρώτων υλών. Μια άλλη πτυχή είναι η οδηγία για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Εγώ τονίσω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας και είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί αυτή η οδηγία μπορεί πραγματικά να δώσει δυνατότητα να κάνουμε μερικά πειράματα καινοτομία τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα στην πολιτική διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα θέματα εξαγωγών <clears throat> νομίζω ότι η οδηγία αυτή θεσπίζει πιο αυστηρές προδιαγραφές οι οποίες όμως θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη. Και απαντώντας και στο ερώτημα της κυρίας Νίμπλα, νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για το ύψος, για το επίπεδο των ε, παρανόμων εξαγωγών. Έχουμε όμως κάποια παράπλευρα στοιχεία για τις διαρροές ουσιαστικά τέτοιων προϊόντων τα οποία εξάγονται με τον τρόπο αυτό και ξέρουμε περίπου 50% πηγαίνουν σε τόπους που δεν είναι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να είναι οι τελικοί. Για τα θέματα της, ε, των παράνομων εξαγωγών έχουμε ήδη, έχω ήδη πει ορισμένα πράγματα. Δεν είναι μονάχα θέμα της ε, εποπτείας στα σύνορα, ξέρουμε ότι πολλές φορές αυτές οι εξαγωγές γίνονται και από οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία και σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Το θέμα τώρα της ανταγωνιστικότητας, της εξόριξης για την ε, Γερμανία και άλλες χώρες δεν μπορώ να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, υπάρχουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση αυτών των περιοχών. Ίσως αν θέλετε μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σε μια έγγραφη υποβολή στην Επιτροπή σας. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω, όπως ε, φαντάζεστε, η γερμανική βιομηχανία ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα των βιομηχανικών ε, πρώτων υλών δεν μας απασχολεί τόσο το θέμα της, ε, των γεωργικών <clears throat> πρώτων υλών. Τώρα, ο κατάλογος των ε, υλικών αυτών θα πρέπει να βασίζεται στην ε, ζήτηση για αυτά τα προϊόντα και στη διαθεσιμότητά τους. Και από τη δική μας πλευρά, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη διαχείριση των σπανίων πόρων είναι πράγματι η αγορά. Φυσικά η πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά, αλλά όχι αποκλειστικά η πολιτική. Υπάρχει χώρος και για την αγορά. Κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την ανακύκλωση είναι ότι χρειαζόμαστε και τους τρεις πυλώνες. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μονάχα σε ένα από τους πυλώνες για να εξασφαλίσουμε την τροφοδοσία της βιομηχανίας με πρώτες ύλες χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα, πέρα από την ανακύκλωση φυσικά, να υπάρξει και η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες που μπορούν να βρεθούν μονάχα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εμπλέκει και την εμπορική μας πολιτική εναντί των χωρών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις εμπειρογνώμονες, λέει ο Πρόεδρος, για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έχουν δώσει και δεχόμαστε και την πρότασή σας να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες, να μας δώσετε μάλλον εσείς περαιτέρω πληροφορίες. Μπορώ να κλείσω λοιπόν αυτό τον πρώτο γύρο της ακρόασης και περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο της ακρόασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούν να έρθουν οι επόμενοι εμπειρογνώμονες στο Προεδρείο, μπορούμε να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Ελάτε κυρίε και κύριοι.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 Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο το, της ακρόασής μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υποφελώς τον χρόνο γιατί έχουμε καθυστερήσει ελαφρά. Ερχόμαστε τώρα στις διεθνείς προοπτικές που είναι το θέμα του δεύτερου πάνελ και θα να καλωσορίσω τους ε, καλεσμένους μας, τον κύριο Έγκερτ, τον κύριο Ντεσά και τον κύριο Σίεμ. Παρακαλώ να με διορθώσετε αν ε, παραμορφώνω τα ονόματά σας και χωρίς να πω πολλά περισσότερα θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Έγκερτ, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντή του Τμήματος οικονομία και Επιχειρήν στο Colorado School of Mines, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις διεθνείς προοπτικές για, την, για τις πρώτες ύλες και την πολιτική πρώτων υλών. Έχετε το λόγο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας να λάβω μέρος σε αυτή την ακρόαση. Λέγομαι Ραντ Έγκερτ, είμαι οικονομολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου στο Conrad School of Mines. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο ασχολείται ιδιαίτερα με τις επιστήμες και τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τη μηχανολογία στις ΗΠΑ. Θέλω να παρουσιάσω μια προσωπική άποψη, μια αμερικανική προσέγγιση και το τονίζω αυτό για να είναι σαφές ότι εγώ δεν σας παρουσιάζω την άποψη της αμερικανικής κυβέρνησης. Είναι η προσωπική μου οπτική γωνία από τις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι η πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης. Σας έχω δώσει ένα έγγραφο κείμενο το οποίο θα σας δοθεί, θα σας διανεμηθεί μετά την ακρόαση, αλλά στα επόμενα λίγα λεπτά θέλω να κάνω μια σύνοψη αυτού του εγγράφου σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι προσωπικού χαρακτήρα αν θέλετε, δηλαδή θα σας παρουσιάσω τέσσερις προτάσεις οι οποίες αντανακλούν την προσωπική μου προκατάληψη αν θέλετε ή την προσωπική μου οπτική γωνία στα θέματα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα το πρωί και το δεύτερο τμήμα θα είναι ουσιαστικά οι άμεσες απαντήσεις στα τέσσερα ερωτήματα τα οποία μου ζητήθηκε να αντιμετωπίσω. Ξεκινώ λοιπόν με τις τέσσερις προσωπικές μου ερωτήσεις, προτάσεις μάλλον η πρώτη μου θέση είναι ότι δεν μας ε, τελειώνουν οι πρώτες ύλε, τουλάχιστον όχι τώρα, το μέλλον. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη ότι ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης για την πρόσβαση στις πρώτες ύλε θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει σπάνης και εξαφανίζονται πια και δεν υπάρχουν πια αυτές οι πρώτες ύλε, κάτι το οποίο είναι μια παρεξήγηση και αυτό με οδηγεί στη δεύτερη θέση την οποία θέλω να τονίσω. Όταν μιλάμε για την διαθεσιμότητα πρώτων υλών ή ορυκτών και την ασφάλεια εφοδιασμού, <clears throat> είναι καλύτερο να σκεφτούμε την γεωγραφία, το χρονικό πλαίσιο και το κόστος. Όταν μιλάμε για κόστος, αναφέρομαι όχι μονάχα για το καθαρά οικονομικό κόστος της εξόρυξης πρώτων υλών και ε, ορυκτών και την ανακύκλωσή τους, που φυσικά ποικίλει από τη μια περιοχή στην άλλη, αλλά και το ευρύτερο λιγότερο ποσοτικοποιημένο κόστος σε επίπεδο περιβάλλοντος και κοινωνικό κόστος που συνδέεται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή. Γεωγραφική πτυχή. Είναι σαφές ότι κάποιες από τις ανησυχίες μας ορίχησαν στη σημερινή ακρόαση αντανακλούν το γεγονός ότι σε για ορισμένα υλικά είναι συγκεντρωμένη γεωγραφικά η παραγωγή τους, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η γεωγραφική συγκέντρωση και η εξάρτηση από τις εισαγωγές όμως δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Μερικές φορές η εξάρτηση από εισαγωγές μπορεί να είναι θετική αν οι εξωτερικές πηγές είναι καλύτερες από τις εγχώριες πηγές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους χρονικούς ορίζοντες, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και του μακροπρόθεσμου επίπεδου. Βραχυπρόθεσμα, το βασικό πρόβλημα με τους ε, βασικούς πόρους της πρώτες ύλες είναι η διαθεσιμότητα και η κίνδυνη να διαταραχθεί αυτή η διαθεσιμότητα. Και το βραχυπρόθεσμο επίπεδο δείχνει ότι οι δυνατότητες παραγωγής εξαρτώνται και από προηγούμενες επενδυτικές αποφάσεις και αποφάσεις προηγούμενες και τρέχουσες των κυβερνήσεων. Αυτά είναι διαφορετικά θέματα από ότι πρέπει να αντιμετωπίσει μια μακροπρόθεσμη προοπτική που έχει να κάνει με τις γεωλογικές συνθήκες, με τις τεχνολογικές ικανότητες και με το ρόλο της δημόσιας πολιτικής για να δημιουργήσει περαιτέρω γνώση στο γεωλογικό επίπεδο και τεχνολογική ικανότητα εξόρυξης. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που θέλω να τονίσω. Το τρίτο είναι το εξής. Ως οικονομολόγος έχω πάντα την τάση να προτιμώ τις λύσεις που δίνει η αγορά και όχι τις λύσεις που δίνουν οι κυβερνήσεις και η ρύθμιση. Επομένως, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι πανάκια η αγορά, δίνει ισχυρά κίνητρα για να υπάρξει καλή διαχείριση των κινδύνων στην ε, απόκτηση πρώτων υλών και στη σωστή χρησιμοποίησή τους. Αν σκεφτούμε την ανησυχία για τις σπάνιε γέες, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μια έκρηξη, μια γενικευμένη ιστερεί, αν θέλετε, η αξόρυξη σε σχέση με τις σπάνιες γιές. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε λίγο χρόνο θα έχουμε πηγές σπανίων γεών εκτός της Κίνας. Οι αγορές επίσης δίνουν σημαντικά κίνητρα για τους χρήστες να εξασφαλιστούν εναντί των κινδύνων που διακρίνουν σε ό,τι αφορά την ε, απόκτηση σημαντικών εισρώων για τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Αυτή η εξασφάλιση λοιπόν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο μπορεί να πάρει και τη μορφή της υποκατάστασης ορισμένων στοιχείων για τα οποία υπάρχει πραγματικά κίνδυνος για την τροφοδοσία. Η τέταρτη θέση την οποία θέλω να τονίσω είναι ότι παρά το γεγονό ότι οι αγορέ είναι ισχυρέ και πάρα πολύ χρήσιμε σε πολλέ περιπτώσει, δεν αποτελούν πανάκια και υπάρχουν <clears throat> επιπλέον και σημαντική ρόλη, ουσιαστική ρόλη που πρέπει να παιχτούν από τι κυβερνήσει και εδώ θέλω να σας πω ποιος είναι, ποιος είναι πιο σημαντική ρόλη που πρέπει να διαδραματίσει μια κυβέρνηση. Καταρχήν να ενθαρρύνουν το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο και αγώνας κατά των περιοριστικών εμπορικών πρακτικών. Δεύτερον, και αυτό πάλι από αμερικανική οπτική γωνία δεν μπορώ να σχολιάσω την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, να βελτιώσουμε την ε, ρυθμιστική διαδικασία έγκρισης και την αποτελεσματικότητά της για εγχώρια παραγωγή ορυκτών και για ανακύκλωση επίσης πρέπει να τονίσω. Να είμαστε προσεκτικοί, εγώ δεν λέω ότι η... πρέπει να υπάρχει προτίμηση στην εξόρυξη και στην ανακύκλωση έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ πιστεύουμε, ότι οι διαδικασίες έγκρισης είναι υπερβολικά επαχθείς και χρονοβόρες. Αναγνωρίζω το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια διαδικασία έγκρισης και προστασία του περιβάλλοντος. Τρίτον, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ρόλος της, για τις κυβερνήσεις στο να ενθαρρύνουν την διάδοση των πληροφοριών, την ανάλυση, την τεχνική και τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη ώστε να έχουμε μια σωστή κατανόηση της κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουμε, να ξέρουμε ποια είναι η φύση του προβλήματος, να έχουμε μια συνετή λήψη αποφάσεων, να έχουμε την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο προεμπορικό στάδιο και συνήθως ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί μόνος του να συλλέξει και να αξιολογήσει όλες αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες. Και όταν μιλάω για πληροφορία, έρευνα και ανάπτυξη, σκέφτομαι για έρευνα που αφορά όλο το κύκλο ζωής των ορυκτών και των ε, πρώτων υλών από την αρχική φάση της εξόρυξης μέχρι την τελική φάση της ανακύκλωσης και ανάκτησής τους. Αυτά είναι λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία που με ενδιαφέρουν για αυτό το θέμα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα τέσσερα ερωτήματα τα οποία μου ζητήσαν να απαντήσω. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπουν οι Ηνωμένε Πολιτείε την τωρινή κατάσταση σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού. όπως και στις ε, ευρωπαϊκές χώρες ίσως δεν υπάρχει καμία ενιαία αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Έχουμε αντιμαχόμενες πολλές φορές απόψεις οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεως και την ε, χάραξη της δημόσιας πολιτικής. Επιπλέον, πρέπει να πω ότι το κίνητρο του να τεθεί σε δημόσια συζήτηση όλη αυτή η προβληματική είναι κάπως διαφορετικό από ό,τι στην Ευρώπη. Η περισσότερη ανησυχία προέρχεται από δύο περιοχές. Καταρχήν, η ανάγκη του να έχουμε την πρόσβαση σε σπάνιες γέες από την Κίνα, που ακούσαμε προηγουμένως σήμερα το πρωί. Και το δεύτερο θέμα είναι η καθαρή ενέργεια. ο ενθουσιασμός που υπάρχει από μια πλευρά για την ηλιακή ενέργεια, την αιωλική ενέργεια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άλλες μορφές καθαρής ενέργειας και τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, που φυσικά όμως χρησιμοποιούν όλες αυτές τις τεχνολογίες μικρές ποσότητες σπανίων στοιχείων, τα περισσότερα από τα οποία δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει σε μεγάλη ποσότητα στο παρελθόν. Υπάρχει λοιπόν το φάσμα της μη διαθεσιμότητας ορισμένων κρισίμων υλικών που θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας. Εκεί λοιπόν υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός για τον τομέα αυτό των εναλλακτικών ενεργειών, παρά το γεγονός ότι στις εφημερίδες πιο πολύ έμφαση έχει δοθεί στην σπάνιδα των σπανίων γεών. Έτσι απαντώ. Νομίζω το πρώτο ερώτημά σας. Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιες είναι οι πολιτικές που, θα, που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμών σε αυτούς τους σπάνιους πόρους. Υπάρχει μια σειρά από πρωτοβουλίε νομοθετικού χαρακτήρα και επίση πρωτοβουλίες της κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μια γενική πολιτική, δεν υπάρχει μια γενική πρωτοβουλία για τις πρώτε ύλε, όπω ε, βλέπω να υπάρχει εδώ στην Ευρώπη. Και δεν είναι απόλυτα σαφή ποιε μορφέ μπορούν να πάρουν αυτέ οι ρυθμίσει στι ΗΠΑ. Αλλά μπορώ να σα συνοψίσω μια σειρά από κέρδιε εξελίξει που έλαβαν χώρα το 2010. Η πρώτη και πιο σημαντική ίσως εξέλιξη έλαβε χώρα στο τέλος του έτους, όταν το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας του Προεδρού δημιούργησε μια υποεπιτροπή για τα κρίσιμα και στρατηγικά υλικά και την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό δεν χτύπησε τα πρωτοσέλιδα, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά το γεγονός ότι αυτή η Επιτροπή δεν έχει ακόμα συνέλθει, θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των πολιτικών σε οριζόντιο επίπεδο σε όλες τις υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Αμερικανικής Κυβέρνησης σε σχέση με τα κρίσιμα και στρατηγικά ε, υλικά που είναι πρώτες ύλες. Είναι λοιπόν μια υποεπιτροπή σε επίπεδο κυβέρνηση που θα έχει εκπροσώπηση όλων των κυβερνητικών φορέων, κυρίω από το Υπουργείο Άμυνα, από το Υπουργείο Ενέργεια, Υπουργείο Ισοτερικών, και φυσικά και από το Φορέα Προστασία του Περιβάλλοντο EPA, και το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνα, NSF. Θα είναι λοιπόν ένα σώμα μέσα από το οποίο η Αμερικανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να διαχειριστεί και να συντονίσει τις πολιτικές στον τομέα αυτό. Δεύτερη σημαντική εξέλιξη στις ΗΠΑ το 2010 προήλθε από το Υπουργείο Ενέργειας. Το Δεκέμβριο ε, έδωσε στη δημοσιότητα τη στρατηγική της για τα κρίσιμα υλικά. που αφορά την δυνατότητα, το φάσμα του να μην υπάρχουν κρίσιμα υλικά τα οποία θα εμποδίσουν την ανάπτυξη καθαρών ενεργειών. Αυτή η στρατηγική λοιπόν η οποία έχει δοθεί σε ένα έγγραφο που βρίσκεται και στο ίντερνετ, το Υπουργείο Έρευνας, ε, Ενεργείας μάλλον, εντόπισε τρεις πυλώνες λίγο διαφορετικούς από τους ευρωπαϊκούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Οι τρεις πυλώνες είναι διαφοροποίηση των αλυσίδων τροφοδοσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον, αναζήτηση υποκαταστάτων για αυτά τα υλικά για τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί η δυσκολία εφοδιασμού και ο κίνδυνη. Και τρίτον, να αυξήσουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Αυτή είναι οι τρει στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Ενέργεια σε σχέση με τα κρίσιμα υλικά. Για τι ε, άμεσε προτεραιότητε, επίση έχει εντοπίσει τρει δράσει για το 2011. Πρώτον, την ανάπτυξη μιας ε, ατζέντα η οποία είναι ολοκληρωμένη για την έρευνα και την ανάπτυξη. Δεύτερον, η αύξηση της ικανότητας του Υπουργείου Ενέργειας για την πληροφορία και την ανάλυση. Πολλοί πιστεύουν ότι η δυσκολία για την σωστή αντίληψη της σημασίας και της σοβαρότητας του προβλήματος τροφοδοσίας προέρχεται από την έλλειψη πληροφοριών. πολλές από τις αγορές για προϊόντα όπως είναι το Ίνδιο, το Τελούριο, το Γάλλιο κτλ. Είναι μικρές αγορές, δεν είναι ιδιαίτερα διαφανείς στον τρόπο λειτουργίας τους. Υπάρχουν μικροί αριθμοί παραγωγών για αυτά τα υλικά και μικροί αριθμοί εταιριών που τα χρησιμοποιούν και πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι οι πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν προβλήματα ανταγωνιστικότητα η μεγάλη διάχυση των πληροφοριών. Επομένω, μια άλλη προτεραιότητα επίση του Υπουργείου Ενέργεια είναι η συνεργασία με διεθνεί εταίρου, ιδίω στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, για να μπορούν να υπάρξουν κοινέ πρωτοβουλίε οι οποίε θα βοηθήσουν να επιλύσουν όλα αυτά τα προβλήματα. <clears throat> αυτά λοιπόν για, τις, ε, για τη στρατηγική του Υπουργείου Ενέργεια. Ένα τρίτο τομέα όπου υπήρξε κίνηση στι ΗΠΑ πέρσι ήταν στον τομέα του διεθνού εμπορίου η κυβέρνηση Ομπάμα διερευνεί ενδεχόμενες παραβιάσεις από την Κίνα των κανόνων του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά προϊόντα που έχουν να κάνουν με την καθαρή ενέργεια. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό το πρόβλημα είναι οι σπάνιες γέες και υπάρχει κατηγορία ότι η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές με στόχο να δώσει προτεραιότητα και πλεονέκτημα στην κινέζικη ε, παραγωγή αγαθών που έχουν να κάνουν με τις καθαρές ενέργειες και για να μπορέσει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούν σπάνιες γένες. Και αυτό έγινε, αυτή η διερεύνηση έγινε μετά από μια λεγόμενη αναφορά 301 βάση του εμπορικού νόμου του 1974 που επιτρέπει σε βιομηχανίες και άτομα να ζητούν από την κυβέρνηση να ξεκινήσει διαδικασίες ε, επίλυση διαφορών στον Παγκοσμίο Οργανισμό Εμπορίου και ήρθε από τη Χαλιβουργία στις ΗΠΑ. Τέλος, το 2010 υπήρξε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες και νομοθετήματα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Όλα αυτά στο στην τελευταία σύνοδο του του Κογκρέσου τελικά δεν οδήγησαν σε τίποτα, αλλά τουλάχιστον ανύψωσαν το επίπεδο της συζήτησης και οδήγησε σε μια δοκιμασία των ιδεών για ενδεχόμενες παρεμβάσεις <clears throat> από την κυβέρνηση στην πολιτική στα θέματα αυτά. Θέλω εδώ να συνοψίσω τις κύριες ιδέες οι οποίες εξήλθανε. Η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, εγγυήσεις δανείων για την εγχώρια παραγωγή κρίσιμων υλικών, μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης για τα περιβαλλοντικά θέματα, καλύτερη πληροφόρηση και ανάλυση, έρευνα και ανάπτυξη και καλύτερη παιδεία και κατάρτιση. <clears throat> Ίσως θα εισαχθούν νέα νομοθετήματα στη νέα σύνοδο του Κογκρέσου που ξεκίνησε στις αρχές του Ιανουαρίου. Τώρα ποια από αυτά τα στοιχεία θα είναι τμήματα της νέας νομοθεσίας, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σαφές, θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Τρίτο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος της επιστήμης και της τεχνολογίας για την προαγωγή των, ε, της ασφάλειας των ε, πόρων. Θα είμαι σύντομος εδώ. Η άποψή μου ως ακαδημαϊκός είναι ότι αυτή είναι η λύση μακροπρόθεσμα για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Όπως σας είπα και πριν, ε, για όλο το κύκλο ζωής από τη γεωλογία μέχρι την διάθεση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Τέλος, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να δουν πώς μπορούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν στον τομέα αυτό. Ε, θεωρώ ότι οι δύο πιο προφανείς ε, περιοχές για συνεργασία είναι η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάλυση τους φυσικά. Οι ε, πληροφορίες θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά, να ληφθούν καλύτερα αποφάσεις για το πώς θα ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις στον τομέα αυτό και δεύτερον συνεργασία στην ε, τεχνική έρευνα και ανάπτυξη και στα δύο μέτωπα ελπίζω να υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχουν ομάδες αν θέλετε εκπροσώπων όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από τους κλάδους και από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αυτές είναι λοιπόν οι προσωπικές μου απόψεις, οι προτάσεις μου και οι απαντήσεις μου στις τέσσερις ερωτήσεις που μου ζητήσατε να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση και τις άλλες παρουσιάσεις που θα ακούσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλό τον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Πάολο Ντεσά, που είναι υπεύθυνο ε, για θέματα φυσικού αερίου, πετρελαίου και πολιτικής, ε, μεταλλευτικής πολιτικής στην Παγκόσμια Τράπεζα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πολύ. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, στον οίκο σας, και να παρουσιάσω τις απόψεις ενός διεθνούς οργανισμού. Θα, θα αλλάξω λίγο το σημείο εστίαση, διότι η Παγκόσμια Τράπεζα δεν εκπροσωπεί καμία συγκεκριμένη κυβέρνηση, ούτε δίνει συγκεκριμένε πληροφορίε για τι ε, πολιτικέ εφοδιασμού των κυβερνήσεων. Ε, Κυρίω εμεί ενδιαφερόμαστε για τι ε, χώρε οι οποίε ε, δεν έχουν πόρου, να τους που έχουν πόρου, να του βοηθήσουμε να έχουν μηχανισμού εκμετάλλευση των εξορρυκτικών του βιομηχανιών. Θα ήθελα να σα δώσω κάποια χαρακτηριστικά του τομέα των πρώτων να σας δείξω γιατί είναι ιδιαίτερος και γιατί χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε θέματα εμπορικών κανόνων και πολιτικών για το τομέα. Ε, ο πρώτος είναι φυσικά η γεωγραφική τοποθεσία. Δεν επενδύουμε στην εξόριξη πρώτων υλών όπου θέλουμε, επενδύουμε εκεί που μπορούμε να τους βρούμε. Οι γεωλογικοί παράγοντες είναι το βασικό κριτήριο για τις επενδύσεις σε πρώτες ύλες. όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις σε πρώτες ύλες. Αυτό δεν γίνεται ε, μόνο με βάση την αποδοτική, ε, τον αποδοτικό καθορισμό και το ε, εργατικό δυναμικό, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες. Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίο μπορεί να έχει πολύ σημαντικά έσοδα και ο καθηγητής προηγουμένω αναφέρθηκε σε δυνατότητες και χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στι χώρες που υπάρχουν ε, μεγάλα αποθέματα ή όπου ανακαλύπτονται αποθέματα και κάποια από αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι πραγματικά κερδοφόρα. Ε, ο ακαδημαϊκός ε, τομέας αναφέρεται σε αυτά ως εισοδήματα. Ε, στην Ινδία, για παράδειγμα, υπάρχει μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με διάφορες δυνάμεις, με παραγωγούς και καταναλωτές για τον τρόπο που καταμερίζεται αυτό το εισόδημα. Φυσικά η έμποροι προσπαθούν να λάβουν την καλύτερη δυνατή τιμή από τους παραγωγούς, αλλά και οι παραγωγοί προσπαθούν να λάβουν όσο καλύτερη τιμή για να πουλήσουν το προϊόν τους. Πάντα λοιπόν υπάρχει αυτή η ένταση για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί αυτό το εισόδημα, αυτό το έσοδο ε, που προκύπτει από την εξόριξη πρώτων υλών. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, αλλά ένα τρίτο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη, κυρίως όσον αφορά την εξόριξη και όχι τόσο το πετρέλαιο, αλλά αφορά και τις δύο πηγές, είναι ότι υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά αποτυπώματα και από περιβαλλοντικής και από κοινωνικής πλευράς. Ε, τα ορυκτά ε, και τα πετρέλαια πολλές φορές επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εξελίξεις. Μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια ε, που έρχονται σε δήμους ή σε περιοχές που έχουν εξορρεκτικές δυνατότητες. Οι επενδύσεις αυτές διαταρέσουν τελείως λοιπόν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στις περιοχές τις οποίες αρχίζουν και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, για το πώς θα καθορίσουμε την εμπορική πολιτική ή μια στρατηγική πρώτων υλών για μεγάλες περιοχές όπως για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού υπησέρχεται τώρα η Παγκόσμια Τράπεζα. Εμείς είμαστε ε, ένας από τους μεγαλύτερους φορείς που δίνουν ε, ε συμβουλές για χάραξη ε, πολιτικής για την εκμετάλλευση πόνου στον αναπτυσσόμενο χώρο. Έχουμε πολιτικές σε πάρα πολλές χώρες και έχουμε βοηθήσει χώρες να αναπτύξουν το ρυθμιστικό και νομικό τους πλαίσιο. Έχουμε καθορίσει ε, ποιοι φορείς είναι αυτοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να εφαρμόσουν το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο. Παρέχουμε δεδομένα και πληροφορίες σε κυβερνήσεις για να τους επιτρέψουμε να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και ε, στο βαθμό που ε, απαιτείται λαμβάνουμε υπόψη και τις τρέχουσες τάσεις και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, των χωρών αυτών για να εκμεταλλευτούν τα ορυκτά τους αποθέματα θέματα και το πετρέλαιο που έχουν με τις μεγάλες, σε συνεργασία με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το ρόλο των διεθνών οργανισμών στον τομέα των φυσικών πόρων Από πλευράς μας θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ε, είναι σε δύο βασικούς τομές. Στον ε, ε, εμπόριο και στην ανάπτυξη. Φυσικά για το εμπόριο ο ΠΟΕ είναι ο βασικός φορέας και αυτοί είναι οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες και επιλύουν τις διαμάχες σε θέματα εμπορίου. Η Παγκόσμια Τράπεζα βέβαια έχει ε, δώσει κάποιες συμβουλές σε χώρες για τις εμπορικές τους πολιτικές ε, και η φυσική πόρη είναι από τα βασικά στοιχεία που δίνουμε στις συμβουλές μας ως προς την πολιτική των χωρών αυτών θέλουμε να μην υπάρχει διάκριση στις πηγές εισοδήματος και οι συμβουλές που δίνουμε είναι για να δημιουργήσουν οι χώρες αυτές ένα ισότιμο πεδίο, όλοι οι επενδυτές να λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση και να βασίζονται στα ίδια κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τους διεθνούς εμπορικούς κανόνες, ε, από τους οργανισμούς, αλλά φυσικά και την εθνική νομοθεσία της, ε, των χωρών που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους. Δεν θέλουμε να έχουμε περιορισμού στην εκμετάλλευση γιατί θεωρούμε ότι μακροπρόθεσμα δεν βοηθούν και βραχυπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσουν ε, εκτείναξη των τιμών ή ε, προβλήματα στη ζήτηση, ε, θέματα τα οποία δεν θεωρούμε, θεωρούμε ότι είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των χωρών παραγωγών. Μία πρόσφατη ανησυχία που έχει ε, προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων είναι η ευμεταβλητότητα των τιμών, η διακύμανση των τιμών. Το πετρέλαιο βέβαια είναι ένα αγαθό το οποίο ε, ενδιαφέρει όλους, αλλά πρόσφατα αλλάζουν οι τιμές των τροφίμων, ε, και τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν πολλούς και αυτό μας έχει δείξει ότι υπάρχει μια τάση να είναι πολύ πιο ε, κειμενόμενες οι τιμές από ό,τι στο παρελθόν. Και εδώ νομίζω ότι πρόκειται και για ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να έχουμε ε, παρέμβαση από πλευράς διεθνών οργανισμών που μπορούν να βοηθήσουν για να αυξηθεί η διαφάνεια των δεδομένων για τις βασικές αγορές πρώτων υλών. Αυτό σχετίζεται και με την παραγωγή, την κατανάλωση και φυσικά με το εμπόριο και τις τάσεις των τιμών. Υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή κάποιες πρωτοβουλίες που συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο G20 μεν, αλλά ε, προάγονται από τις ευρωπαϊκές ε, χώρες για να αυξηθούν οι πληροφορίες και το επίπεδο διαφάνειας για τις αγορές των βασικών αγαθών. Και εδώ θεωρούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς ε, με τις συμβουλές μας. Η βασική μας ανησυχία τώρα για τους φυσικούς πόρους είναι από πλευράς ανάπτυξης. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη γιατί θεωρούμε ότι η ανάπτυξη των εξορρυκτικών βιομηχανιών θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη ε, των χωρών που είναι πλούσιες σε φυσικές ε, πόρους σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν στην Παγκόσμια Τράπεζα έχουμε έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και πόρους στην έρευνα ε, προσπαθώντας να, να καταδείξουμε με ποιο τρόπο μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά η ανάπτυξη των φυσικών πόρων και της εξορρυκτικής βιομηχανίας στο βιωτικό επίπεδο των χωρών που έχουν φυσικούς πόρους και φυσικά υπό ποιες συνθήκες θα μπορέσουν αυτά τα τρέχοντα φαινόμενα της μείωσης ε, ε, και της έλλειψης κάποιων προϊόντων να αντιμετωπιστεί. Δεν θεωρούμε ότι αποτελεί κατάρα ε, για τις χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικές πόρες. Θεωρούμε ότι ε, αν τους δοθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αυτός ο φυσικός πλούτος μπορεί να ε, μετατραπεί σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και θεωρούμε ότι είναι βασικός ο ρόλος που μπορούμε να διαδραματώσουμε εμείς, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να κάνουν αυτή τη μετατροπή. Υπάρχουν πέντε τομείς στους οποίους επικεντρώνουμε την προσοχή μας και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι προκειμένου οι χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικές πόρους να αυξήσουν το φυσικό τους πλόητο και να γίνει αυτό βιώσιμη ανάπτυξη. Και εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας για τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες από τις χώρες ε, ε εισαγωγής ε, και εδώ νομίζω ότι εμπίπτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυτικέ χώρες λοιπόν οι οποίες εισάγουν προϊόντα ε, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις τιμές και θεωρούν ότι ο βασικός είναι ο, βασικός δείκτης αποδοτικότητας για τον εφοδιασμό. Ε, από το 2004 όμως η ταχύτερη ανάπτυξη ε, των BRICS των αναπτυσσόμενων χωρών με μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης και υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης μας έχει ε, δώσει νέες τάσεις και έχει δημιουργηθεί ένας νέος ανταγωνισμός ε, για την πρόσβαση σε πόρους. Κάποιες από αυτές τις χώρες BRICS έχουν καταφέρει με πολύ έξυπνο τρόπο να διαμορφώσουν το ρόλο των, ε, ε, της εμπορίας των υλικών. Έχουν αλλάξει το διεθνές προσκήνιο στις επενδύσεις σε πρώτες ύλες και στο εμπόριο πρώτων υλών και έχουν καταφέρει μέσω των εμπορικών τους πολιτικών να κάνουν το μειονέκτημά τους πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός υποδομών και πόρων, η δυνατότητα να επεκταθούν ε, σημαντικά ποσά σε δάνεια, ε, υπό τη μορφή δανείων για υποδομές, τα οποία ε, υποστηρίζονται και διασφαλίζονται από την ανάπτυξη των πρώτων υλών τους. Η πρότασή μου λοιπόν για τους παραδοσιακούς ε, παίκτες και εισαγωγές, εισαγωγής πρώτων υλών είναι ότι υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθούν λίγο οι παραδοσιακές πολιτικές εφοδιασμού τους, να λάβουν υπόψη τι νέες τάσεις στην αγορά και τον νέο ανταγωνισμό από τις χώρες BRICS. Όπως σα έλεγα, ε, το βασικό στοιχείο γι' αυτό από πλευράς ε, Παγκόσμιας Τράπεζας είναι να αναπτύξουμε ενεργές πολιτικές συνεργασίες με τις ε, χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικές πόρους και για να παραφράσω μια παραδοσιακή έκφραση που χρησιμοποιούν συχνά οι Κινέζοι, για να έχουμε προτάσεις win-win που θα είναι υποφελής όχι μόνο για τη χώρα η οποία κάνει τις αγωγές, αλλά θα έχουμε και ε, βιώσιμη ανάπτυξη για τις χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια στρατηγική για τις πρώτες ύλε, ε, για τις χώρες που κάνουν αγωγές όπως είναι η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στις ε, εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν είναι μόνο θέμα του πώς έχω πρόσβαση εγώ στις πρώτες ύλες αλλά πώς θα σας μπορέσω να σας βοηθήσω να αναπτύξετε τις, ε, την εκμετάλλευση των πρώτων υλών σας κατά τρόπον ώστε να οπεφοληθώ εγώ, γιατί θα μπορείτε να τροφοδοτείτε την δική μου βιομηχανία, αλλά θα υποφοληθείτε κι εσείς, γιατί αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων σας, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στο πληθυσμό και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η ενσωμάτωση των πολιτικών πολιτικών ε, τροφοδοσίας ε, για τις ε, χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικές πόρους είναι για μας το κλειδί της επιτυχίας στις νέες πολιτικές εφοδιασμού. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς είναι το θέμα της διαφάνειας. Η διαφάνεια μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την ε, ε, καλή λειτουργία των ε, αγορών, διότι η έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο έχουν ήδη αναλυφθεί κάποιες πρωτοβουλίες και ελπίζουμε ότι μία αποτελεσματική ε, στρατηγική εφοδιασμού θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες είναι υπέρ της αύξηση της διαφάνειας της αγορές πρώτων υλών. Τρίτον, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι πρώτες ύλε, ιδίως από το 2004 και μετά, είναι μια πολύ ε, επικερδής ε, βιομηχανία και οι χώρες εισαγωγής θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η χώρα που κάνει την εξαγωγή των πρώτων υλών θα πρέπει ε, να αποζημιώνεται καταλήλως ε, για τα ύλε που εξάγει. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερα φορολογικά καθεστώτα για τις χώρες που κάνουν εξαγωγές ε, πρώτων υλών αυτό είναι όλο ένα και πιο σημαντικό στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στις ε, πολιτικές συνεργασίες μεταξύ ε, χωρών εισαγωγής και χωρών εφοδιασμού και φυσικά θα πρέπει να αναγνωρίζετε ότι η κατάλληλη ε, αποζημίωση για τους πόρους αυτούς θα πρέπει να αποτελεί κανεί και αναγκαία συνθήκη για τη συνεργασία η καταβολή φυσικά των φόρων και η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, ιδίως σε χώρες όπου τα θεσμικά όργανα δεν είναι πολύ ε, ισχυρά. Ε, πολλές φορές ε, προσεγγίζονται αυτές οι χώρες και ζητούνται, ζητείται προτιμησιακό καθεστώς και καλύτερη πρόσβαση ε, στις πρώτες ύλε και τους γίνεται μια προσφερά η οποία δεν είναι και καλύτερη δυνατή για την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Καλύτερη λοιπόν πληρωμή για τις χώρες αυτές και μια καλύτερη στρατηγική. Το τέταρτο στοιχείο είναι λίγο ακαθόδες για τις ε, χώρες εισαγωγές, διότι πάντα οι χώρες ε, θέλουν να έχουν περισσότερη αξία για τα προϊόντα τους και αυτό φυσικά δεν συνάδει με την αναπτυξιακή πολιτική ε, των χωρών που χρειάζονται πρώτες ύλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε απαραίτητο μείωση, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε για τις χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε πόρους είναι ότι ε, υπάρχουν δυνατότητες για να δημιουργηθούν ε, ομάδες ε, ε, ανθρώπων που μπορούν ε, να παρέχουν ε, υπηρεσίες και αγαθά, να συμμετέχουν στα προγράμματα της εξορρυκτικής βιομηχανίας. Για παράδειγμα, η Χιλή και η Ποτσουάνα, για να σας δώσω και ένα παράδειγμα από την Αφρική, κατάφεραν να αναπτύξουν καταλήλως τη βιομηχανία. Υπάρχει θετική ανάπτυξη. Έχουμε πλέον στοιχεία ε, ε, που δείχνουν ότι αναπτύσσονται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες τους. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό λοιπόν παράγοντα, τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη, διότι συνεισφέρει ε, στην πιο σημαντική φιλοδοξία μιας χώρας που κάνει εξαγωγές. Τέλος, μια τελευταία παρατήρηση, το ανέφερα και στην αρχή, είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις τοπικές κοινότητες. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο μια αποτελεσματική εμπορική πολιτική ε, και να έχουμε κατάλληλες τιμές για την τράπεζα, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες που είναι αυτές οι οποίες ε, ε, επηρεάζονται άμεσα από μια εξέλιξη στη χρήση των πόρων τους, είναι αυτές οι οποίες θα αναπτυχθούν καλύτερα σε χώρες της Λατινική Αμερική διαπιστώνουμε όλο ένα και περισσότερο ότι ε, δημιουργούνται διαμάχες. Ε, στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, σοβαρές αντιρρήσεις για την ανάπτυξη των πετρελαϊκών προγραμμάτων, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα αντάλλαγμα οι ίδιοι και θα πρέπει να τους προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα είναι επιφελείς για αυτούς. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, ποια μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να ε, παγιώσουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις πολιτικές για τις πρώτες ύλε. Τα περισσότερα τα έχουμε ήδη αναφέρει επανειλημμένως. Να υπενθυμίσω κάποια από τα πιο προφανή. Καταρχάς πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, των χωρών που είναι πλούσιοι σε φυσικές πόρους για να κάνουν καλές συμφωνίες για τις πρώτες ύλες, διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, είναι όλο ένα και πιο περίπλοκες οι συμφωνίες οι οποίες επιτυγχάνονται με τις ε, κυβερνήσεις, ε, υπάρχουν θέματα υποδομών, επενδύσεων σε αγορές, σε πιο προηγμένες ε, οικονομικές τεχνικές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι κυβερνήσεις και οι χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικές πόρους κατανοούν τι κάνουν και να μπορούν να λαμβάνουν καταλληλότερες αποφάσεις. Εδώ λοιπόν και η Παγκόσμια ε, Τράπεζα αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμών όπως για παράδειγμα η Αναπτυξιακή Τράπεζα επενδύουν και διασφαλίζουν ότι όταν οι κυβερνήσεις αποφασίζουν για την ανάπτυξη και χρήση των πρώτων υλών τους και υπογράφουν συμφωνίες με επενδυτές γνωρίζουν καλά τι κάνουν και οι αποφασίσει λαμβάνονται με διάφορο τρόπο. Δεύτερον, οι κυβερνήσει πρέπει να γνωρίζουν τι διαπραγματεύονται. Οι εμπορικέ πολιτικές για τις πρώτε ύλε προς το παρόν χαρακτηρίζονται από την ε, λεγόμενη πληθώρα πληροφοριών. Αφενός υπάρχει μια επιχείρηση, κάποιος επενδυτής ή κάποιος εμπορευόμενος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και γνωρίζει πολύ καλά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της χώρας ε, και τα αποθέματα ε, στα οποία θέλει να επενδύσει και από την άλλη υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες έχουν ελάχιστες πληροφορίες ε, για τον φυσικό τους πλούτο, τη φυσική τους κληρονομιά. Και αυτό λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός ε, ε, τομέας για δυνητική συνεργασία, να υπάρχουν ε, γεωλογικές πληροφορίες για χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους και εδώ πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια των πληροφοριών για τις αγορές πρώτων εμιλών. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, νομίζω ότι κράτησα το καλύτερο για το τέλος, για να ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχει διαφάνεια στις αγορές και υπάρχουν καλές συμφωνίες για τις κυβερνήσεις, ένα σημαντικό στοιχείο είναι να είναι υπόλογες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι οργανώσει τη κοινωνία των παλετών σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρου, αλλά και σε χώρες εισαγωγή, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και πρωτίστω οι κυβερνήσεις να είναι υπόλογε για τι αποφάσεις που λαμβάνουν. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Σεάμ που είναι αναπληρωτής διευθυντής για θέματα ασφάλειας των τροφίμων και οικονομικής ανάπτυξης ε, στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων ε, και Εξωτερικών Υποθέσεων στη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έρευνα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρουσιάσω την γαλλική προσέγγιση στο G20 σε σχέση με τα θέματα πρώτων υλών. Θα ήθελα καταρχήν να υπενθυμίσω ότι οι πρώτες ύλες και ιδιαίτερα το θέμα της διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας του G20. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να το υπενθυμίσει μόλις προχτές τη Δευτέρα κατά την συνέντευξη τύπου κατά την έναρξη της Προεδρίας του G20 και του G8 από τη Γαλλία. Γιατί ναι. αποτελεί για μας προτεραιότητα το θέμα. Κάνουμε την εξής διαπίστωση. Καταρχήν, στην αγορά πρώτων υλών υπάρχουν εντάσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και με τις προοπτικές ε, που υπάρχουν, ε, οι προοπτικές είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση ενώ παραμένει μακροπρόθεσμα περιορισμένη η προσφορά και θα καταλήξουμε σε ε, μία οικονομικοποίηση της αγοράς των πρώτων υλών μακροπρόθεσμα και αυτό οδηγεί σε αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών των πρώτων υλών. Και αυτή η μεταβλητότητα των τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί στην αποσύνδεση της εξέλιξης των τιμών από τα βασικά στοιχεία της αγοράς, την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διαμόρφωση αποθεμάτων γιατί αποτελεί κατάλληλο χώρο το G20 για τα θέματα αυτά. Διότι το G20 συγκεντρώνει τις πιο σημαντικές οικονομίες του κόσμου, τους βασικούς φορείς της αγοράς και των πρώτων υλών. Οι δράσεις του G20 στο θέμα αυτό ξεκίνησαν πολύ πριν τη Γαλλική Προεδρία του G20 και θέματα διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών υπάρχουν ε, ήδη ε, στο G20 του Πίτσπουργκ ε, ή του Τορόντο ή της Σεούλ. Θα χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα σας πω τι προτείνουμε να κάνουμε για τις οικονομικές αγορές πρώτων υλών και το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθεί με την προσέγγιση μας για την πραγματική αγορά των πρώτων υλών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ενεργειακές πρώτες ύλες και στις γεωργικές πρώτες ύλες, γιατί σε αυτά τα θέματα θα είναι πιο διαρθρωμένη η προσέγγιση του G20. Καταρχήν για τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εδώ και καιρό είναι αντικείμενο στο οποίο εργάζεται το G20 και επί Γαλλικής Προεδρίας θα ασχοληθούμε με τα συμπεράσματα της Σεούλ από τον Νοέμβριο του 2010 όπου δόθηκε μια εντολή στην Διεθνή Επιτροπή στην Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Χρεογράφων για να ασχοληθούν με τα παράγωγα προϊόντα για τις ε, Πρώτε ύλε, ούτω ώστε τον Απρίλιο του 2011 να ε, είναι έτοιμη μια έκθεση που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε την κερδοσκοπία γιατί θα ήταν αδύνατο να επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο. Στόχο μα είναι να δούμε ποιε είναι οι γενικέ αρχέ τις οποίες θα πρέπει να δεσμευθούν να τηρούν οι εταίροι του G20 στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, για τα παράγωγα προϊόντα των εμπορευμάτων. Οι βασικές αρχές είναι η διαφάνεια, διαφάνεια ε, των ε, συναλλαγών, ούτως ώστε να είναι γνωστές όλες οι κινήσεις στην αγορά παραγόγων προϊόντων. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές συναλλαγές χωρίς να είναι εμφανείς και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα. Είναι over the counter συναλλαγές και θέλουμε να έχουμε καλύτερη διαφάνεια για τις συναλλαγές αυτές. Ακόμη θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους φορείς, τους οργανισμούς που εκτελούν τέτοιες συναλλαγές, για να έχουμε κάποιο εργαλείο που θα μας επιτρέψει μακροπρόθεσμα να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών εμπορευομένων δηλαδή αυτών που ε, οι ίδιοι ασχολούνται με τα προϊόντα και αυτών που έχουν μόνο ε, οικονομικό κέρδος ως στόχο. Δεν θέλουμε να υπάρξουν στην αγορά υπερβολές που ε, θα διαβρώσουν το μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών. Και τέλος θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις πραγματικές αγορές εμπορευμάτων. Αυτή η δουλειά στις χρηματοοικονομικές αγορές θα ολοκληρωθεί με μία έκθεση μια εκθεση μιας μελέτης που θα υποβάλει στους Υπουργούς Οικονομικών του G20 για να διευκρινίσει τους όρους και τις συνέπειες ε, της ε, διακύμασης των τιμών και μακροοικονομικά τις συνέπειες επί του πληθωρισμού και επί του ισοζυγίου πληρωμών. Το δεύτερο τμήμα τη παρέμβασή μου είναι αυτά τα οποία προτείνουμε να κάνουμε στις πραγματικές αγορές προϊόντων και εμπορευμάτων, ξεκινώντας από την ενέργεια διότι οι εργασίε του G20 για την ενέργεια έχουν ήδη ξεκινήσει και εμείς θα συνεχίσουμε επί γαλλική προεδρία τι εργασίε αυτές. Σα υπενθυμίζω ότι αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει το G20 είναι να βελτιώσει την διαφάνεια της πληροφόρησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Τζοντάι για ε, την βελτίωση ε, της πληροφόρησης ε, στις αγορές και για να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και για τα αποθέματα και για τις επενδύσεις του πετρελαϊκού κλάδου. Πέρα από την διαφάνεια της πληροφόρησης, η ομάδα ενέργειας του G20 εργάζεται και για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Στηριζόμαστε και στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και στο Διεθνές Φόρουμ για την Ενέργεια. Προτείναμε στους εταίρους μας, πέρα από τα δύο αυτά βασικά θέματα, διαφάνεια και ε, σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, να αρχίσουμε και κάποιες εργασίες ε, για την καθαρή ενέργεια και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Για τις γεωργικές και διατροφικές πρώτες ύλες, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας νέος τομέας. Το G20 έχει με ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, αλλά ποτέ δεν δούλεψε λεπτομερώς πάνω στον τρόπο μείωσης της μεταβλητότητας των τιμών και μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων ε, στις πιο, στα πιο ευάλωτα προϊόντα. Στον τομέα αυτό λοιπόν θα δουλέψουμε πάνω στο σχέδιο δράσης της ΣΕΟΥΛ για την ανάπτυξη ένα σχέδιο δράσης το οποίο έδωσε εντολή σε οκτώ διεθνείς οργανισμούς να υποβάλουν μία έκθεση περίπου κατά τα τέλη Μαρτίου. Οι οκτώ αυτοί διεθνείς οργανισμοί είναι ο Οργανισμός ε, για τη Γεωργία και τη Διατροφή ΦΑΟ, το Διεθνές Διατροφικό Πρόβλημα, το Διεθνές ε, Πρόγραμμα Γεωργικής Ανάπτυξης, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δόθηκε λοιπόν αυτή η εντολή μέσα στο πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των τροφίμων και η Γαλλική Προεδρία του G20 πρότεινε στους εταίρους να οργανωθεί μια συνάντηση Υπουργών Γεωργίας του G20 κατά τα τέλη Ιουνίου για να ασχοληθεί με το θέμα της μεταβλητότητας των τιμών ε, στον τομέα των ε, γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Δεν θα σας εκπλήξω αναφέροντάς σας τα βασικά θέματα πάνω στα οποία θέλουμε να δουλέψουμε. Τα βασικά θέματα είναι η διαφάνεια, η διεθνή συνεργασία και συντονισμός, ούτω ώστε να ασχοληθούμε με τα θέματα περιορισμού των εξαγωγών και πολιτικών αποθεματοποίησης ένα τρίτο θέμα είναι τα μέσα κάλυψης και διασφάλισης των πιο ευάλωτων προϊόντων. Και τέταρτο θέμα, η αύξηση της παραγωγής ή η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγικότητας σε σύνδεση με υπεύθυνες πρακτικές γεωργικών επενδύσεων. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι για τα θέματα αυτά η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί. Συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων του G20. Είναι σχετικά νέο το θέμα αυτό και οι κανόνες εργασίας μέσα στο G20 απαιτούν την ομοφωνία και τη συνένεση. Δεν προωθούνται ανταγωνιστικές θέσεις, αντιθέτως θέλουμε να αναζητήσουμε στοιχεία συνένεσης και συμφωνίας τα θέματα των ορυκτών πρώτων υλών, των πρώτων υλών ε, που δεν είναι στον ενεργειακό τομέα και στη γεωργία, δεν αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένων εργασιών. Παρ' όλα αυτά, αυτά που μπορούμε να κάνουμε ε, για, τα, ε, για τον τομέα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και για τα εμπορεύματα θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τη διεθνή συνεργασία, ε, ούτως ώστε να υπάρξει σωστή αντίδραση για το θέμα της μεταβλητότητας των τιμών των πρώτων υλών. Και βασιζόμαστε στη συνεργασία με όλους τους εταίρους, ιδίως όμως με τους Ευρωπαίους εταίρους, διότι τα στοιχεία ε, επί των οποίων σας είπα ότι θα εργαστούμε, αντιστοιχούν απολύτως στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό όπως παρουσιάζεται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, την οποία με ανυπομονησία αναμένουμε στην αναθεωρημένη εκδοχή της μέσα στις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ακούσει λοιπόν πολλές πρόσθετες πληροφορίες από ε, τους ε, ομιλητές μας. Ο κύριος Παλτσίτης είναι ο πρώτος ομιλητής ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις πλήρες πληροφορίες που μας έχουν δώσει σε σχέση με τα θέματα των πρώτων υλών και οίκοθε εννοείται ότι η σημερινή συζήτηση θα επηρεάσει και την ε, χάραξη της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος καθηγητής Ντεσά τόνισε ότι δεν πρέπει μονάχα να μας ενδιαφέρει η απόκτηση των πρώτων υλών, αλλά η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο καταδεικνύει ότι τα υλικά αυτά τα οποία εισάγονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο και αντιμετωπίζουμε μία σειρά από χώρες οι οποίες παράγουν αυτά τα, αυτές τις πρώτες και οι οποίες πλήττονται από πολιτική αστάθεια και αυτό φυσικά οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών η αυξήση των τιμών λοιπόν στις χώρες αυτές είχε πραγματικά κάποια συνάφεια με την πολιτική αστάθεια. Μήπως μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η πολιτική κατάσταση σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να <clears throat> αντιμετωπιστεί ως επηρεάζουσα την εξόριξη αυτών των υλικών. Πολύ πρόσφατα έχουν υπογράψει μεγάλες εταιρείες εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως αυτές που ανέφερα και έχουν εισαγάγει πρώτε ύλε από τις χώρες αυτές, αλλά ισχύει εξίσου το ότι όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν γίνει με έναν τρόπο αδιαφανή και τα χρήματα τα οποία επενδύονται και δαπανώνται στην Αφρική και στην Ασία συγχρόνως <clears throat> χρηματοδοτούν και τροφοδοτούν εγκληματικές ενέργειες. Να επανέλθω λοιπόν σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν στην ε, Κίνα. ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών έρχονται από την Κίνα και ελέγχονται από τις κινέζικες αρχές. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι χώρες εταίροι μας θα μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι συνθήκες εμπορίου υπόκεινται σε πολύ αυστηρότερη κανονιστική ρύθμιση. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Πολιτείες μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και αυτό φυσικά θα συμβάλλει στην σταθερότητα των χωρών αυτών που εξάγουν αυτές τις πρώτες ύλες. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρία Ουλσκοκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συζητητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον το να ακούσουμε ποιος είναι ο, ρόλος και τις Παγκόσμιας Τράπεζας και επίσης ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για την ισορροπία μεταξύ των παραγωγών και των <clears throat> καταναλωτών των πρώτων αυτών υλών. Έχω να θέσω δύο ερωτήματα. Τα αγροτικά, οι αγροτικές πρώτες ύλες και αυτές έχουν έρθει στο προσκήνιο πρόσφατα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα λόγω της αύξησης των τιμών. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική αβεβαιότητα για τα θέματα αυτά. Όταν μιλάμε λοιπόν για στρατηγικά υλικά, μήπως θα έπρεπε να σκεφτόμαστε αυτόματα και τα... τις αγροτικές πρωτεσίλες, τα βασικά προϊόντα στη γεωργία. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι πρόσφορο να μιλάμε μονάχα με την έννοια της πρώτης ύλη. Είναι πολύ σημαντικό προφανώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουμε μια στρατηγική πρώτων υλών. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να την αναπτύξουμε σε ένα ευρύ επίπεδο Νομίζω ότι στην περίπτωση όμως των γεωργικών βασικών προϊόντων η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει περισσότερο με τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον γεωργικό τομέα. Και ίσω αυτό μπορεί να ισχύει σε κάποιο βαθμό και με τι άλλε πρώτε ύλε και την ενέργεια. Μήπω θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μα περισσότερο στι άλλε πτυχέ που δεν έχουν να κάνουν με τα γεωργικά θέματα. Και τώρα το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να κινηθούμε στον τομέα των πρώτων υλών, τουλάχιστον σε τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσαμε για την ε, Κίνα και την Αφρική. Αλλά έχουμε και ένα νέο χώρο από τον οποίο μπορούν να προέρχονται τέτοιε κέρυε πρώτε ύλε. Είναι η περιοχή του, της Ακτικής όπου υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν συνομιλίες, συμφωνίες μεταξύ διαφόρων εταίρων. Μήπως μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το χώρο της Ακτικής από ό,τι έχει καταστεί δυνατόν να πετύχουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου όπου υπήρξε μια εκμετάλλευση, μια απόλυτη και χωρίς όρια εκμετάλλευση των πόρων εκεί. <coughs> Αυτό το ερώτημα θα ήθελα να το θέσω τώρα στον κύριο Έγκερτ, καθηγητή κύριο Έγκερτ. Είπατε ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη γαλήνη σε σχέση με το θέμα της σπάνιδος των ε, πρώτων υλών. Πώ καταλήγετε σε αυτό το συμπέρασμα. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε τελικά και καλύτερα ποια είναι τα, οι αιτίε που σα οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα και ποια πορίσματα μπορείτε να εξάγετε από αυτό. Γιατί αυτό φυσικά επηρεάζει πάρα πολλά από αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί. Και μετά ο κύριος Κόφερ ήθελε να λάβει το λόγο και βγήκε για κάποια στιγμή και ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο γύρο απαντήσεων και ξεκινάμε τον κύριο Ζήμου η Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με το προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει βεβαίως. Αυτή είναι και η προσέγγιση των G20 γιατί έχουμε αντιμετωπίσει τρία θέματα τις αγορές κινητών αξιών που δεν κάνουν ιδιαίτερη διάκριση σε σχέση με τα προϊόντα και χωριστά τις αγροτικές αγορές όπου χρειάζεται να μιλήσουμε με τους ειδικού στα θέματα ε, τροφιμικής ασφάλειας και από την άλλη μεριά την ενεργειακή αγορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφοροποίηση, βεβαίω χρειαζόμαστε. Αυτέ είναι οι αρχέ επί των οποίων εστιαζόμαστε. Ο διάλογο μεταξύ παραγωγού και καταναλωτήου, η διαφάνεια και η ενισχυμένη συνεργασία. Όλα αυτά είναι βασικέ αρχέ οι οποίε εφαρμόζονται συμπούρμπουλα και συλλήγουν σε όλε αυτέ τι αγορέ. Η Ακτική δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει στο G20 μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. το, στον κύριο Ζάθε, Σάθε να λόγο. Από την Παγκόσμια Τράπεζα θέλετε να απαντήσετε κάποιο ερώτημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα μικρό σχόλιο για την σπάνιδα των πρώτων υλών. Συμφωνώ με τον κύριο Έγκετ, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν υπάρχει σπάνης, ακόμα και η βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχουμε μεγάλες εντάσεις σε συγκεκριμένες αγορές είναι ένα πολύπλοκο θέμα αυτό, όχι τόσο επειδή επηρεάζεται από την πολιτική αστάθεια. Πολλές φορές ο καιρός παίζει ένα σημαντικό ρόλο και οδηγεί σε μεγάλες ε, διαταραχές της, ε, του εφαρμοσμού της αγοράς. Η Αρκτική είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θεωρούμε ότι η Αρκτική είναι ένα είδος καταφυγίου, φυσικού καταφυγίου, όπου η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να υπερισχύσει τι ανάπτυξη των φυσικών πόρων που περικλεί η Αρκτική. Και υπάρχει φυσικά η ένταση μεταξύ της εκμετάλλευσης και της ε, ανάπτυξης μιας ε, διεθνούς ε, σύμβασης για να προστατευτεί αυτή η περιοχή. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση λοιπόν για το θέμα της ακτικής. Ευχαριστώ. Και ο καθηγητής Έγκερτ. Να απαντήσω στην πρόκληση που μου απίθυνε ο πρόεδρος σας. Μήπως είμαι υπερβολικά χαλαρός σε σχέση με την ύπαρξη και διαθεσιμότητα φυσικών πόρων. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Όταν μιλάω για διαθεσιμότητα πρώτων υλών, υπάρχουν τέσσερις ή πέντε συντελεστές αυτής της διαθεσιμότητας. Γεωλογική διάσταση, αν υπάρχει στο φλοιό της γης αυτός ο φυσικός πόρος, υπάρχει τεχνική διάσταση, αν υπάρχει αυτός ο πόρος, έχουμε την τεχνολογία εξόριξης <clears throat> και επεξεργασίας αυτού του φυσικού πόρου. Υπάρχει μια ευρεία διάσταση που είναι κοινωνική, ε, περιβαλλοντική και γεωπολιτική αν θέλετε. Το θέμα του αν μπορούμε να εξορίξουμε αυτές τις πρώτες με έναν τρόπο ο οποίος συνάδει με, τις την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του περιβάλλοντος μπορούμε να τον εξορίξουμε αυτόν τον πόρο με τρόπους οι οποίοι συνδέονται με τις με τη θέληση και την προτίμηση των τοπικών κοινοτήτων όπου λαμβάνει χώρα η εξόριξη αυτή. Επίσης είναι διαθέσιμος αυτός ο πόρος με έναν τρόπο που είναι συμβατός με την εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε. Και τέλος υπάρχει και η οικονομική διάσταση της διαθεσιμότητας. Μπορούμε να βρούμε αυτόν τον πόρο, να τον εξαγάγουμε, να τον εξορίξουμε, να τον εκμεταλλευτούμε με έναν τρόπο που είναι αποδεκτός σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και συγχρόνως αποκομίζοντας κάποιο κέρδος και με οικονομικά κίνητρα για να το κάνουμε αυτό. Εγώ αυτό θέλω να πω λοιπόν είναι ότι γενικά ο πιο ουσιαστικός περιορισμός δεν είναι το αν υπάρχει στο φλοιό της γης ένας πόρος ή όχι, γιατί οι άλλες διαστάσεις μπορεί να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο είναι πιο σημαντική περιορισμοί, τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας δώσω ω απάντηση σε αυτό το ερώτημα και μπορώ να σταματήσω εδώ αν θέλετε. Για την Αρκτική δεν μπορώ να κάνω σχόλια. Υπήρξε το ερώτημα του αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερφιλόδοξη ή ακολουθεί μια πολύ πολυμέτωπη πολιτική προσπαθώντας να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα, τα κρίσιμα και στρατηγικά στοιχεία πρώτων υλών, αγροτικά προϊόντα, διακύμανση τιμών, όλα αυτά μέσα σε μια συνολική πολιτική κατεύθυνση. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει ένα φάσμα θεμάτων που έχουν διαφορετική φύση. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά συλλήβδεν με μια κοινή πολιτική. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο έχω να σε εκθέσω μια άποψη. Και σταματάω εδώ. Κύριος Μπιουτικόφερ έχει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω ερωτήσει προ όλου ε, του ομιλητέ. Προ τον κύριο Έγκερτ, καταρχήν. Καθηγητά, κύριε Έγκερτ. Ο εκπρόσωπο εμπορίου των Ηνωμένων ε, Πολιτειών δεν ε, συμφώνησε με το αίτημα ε, των εργαζομένων από τον, τομέα του Χάλιβα και θα ήθελα να μου πείτε πώς το ερμηνεύετε εσείς. Ε, ήταν μια διπλωματική αντιμετώπιση για να μην υπάρξουν διενέξεις στο πλαίσιο μιας διαδικασίας του ΠΟΕ ή δόθηκαν διασφαλίσεις από τους Κινέζους ε, προς ε, την Υπουργό Εξωτερικών, κυρία Κλίντον, ή εξετάζεται περαιτέρω το θέμα. Έχω επίσης και μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ντεσά. Μιλήσατε πολύ για τη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια, όπως η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στην εξωτερική βιομηχανία, όπως επίσης και το Say What You Pay. Υπάρχουν δηλαδή πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια. Και στο πλαίσιο της νομοθεσίας Dodd Frank στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν στην χρηματοοικονομική αγορά υπάρχουν διατάξεις για τη διαφάνεια, για τα κρίσιμα υλικά. Υλικά που ενδέχεται να προκύπτουν από περιοχές όπου υπάρχει εμφύλιος πόλεμος κλπ. Θεωρείτε ότι είναι θετική αυτή η προσέγγιση και υποστηρίζετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και για τον κύριο Έγκερτ και πάλι μια ερώτηση για το συγκεκριμένο αυτό θέμα της νομοθεσίας Dot Frank προχωρεί η διαδικασία ε, και μια ερώτηση προς τον κύριο Σεάμ σχετικά με την κερδοσκοπία. Είπατε ότι θέλετε να αντιμετωπίσετε την κερδοσκοπία και ε, ε, γι' αυτό θα δοθεί η δυνατότητα και μέσω της διαφάνειας να γνωρίζουμε ποιος εμπλέκεται. Υπάρχει μια προσπάθεια και στις ΗΠΑ μέσω της νομοθεσίας και από τα σχόλια που έχω διαβάσει δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό αυτό το μέσον. Εσείς ε, τι περαιτέρω βήματα έχετε κατά νου να λάβετε για να το αντιμετωπίσετε. Και μια δεύτερη ερώτηση. Η Γαλλική Προεδρία του G20 θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα της κερδοσκοπίας ε, στα είδη διατροφής. Ε, εσείς βλέπετε να υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της κερδοσκοπίας με τις βιομηχανικές πρώτες ύλες ή θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό το θέμα της κερδοσκοπίας ε, σε άλλες ύλες εκτός από τις ε, βιομηχανικές και πώς πώ εξηγείται τι προτεραιότητε τη Γαλλική Προεδρία και μήπω τα οποία η Γαλλική υλε εκτος απο τις βιομηχανικες και πως εξηγειτε τις προτεραιοτητες της θέλει να θεσπίσει για να αντιμετωπίσει την κερδοσκοπία ε, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων αργότερα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα βιομηχανικά προϊόντα. ακόμη νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη το να χρησιμοποιήσουμε την ε, ε, ασύμμετρη την αντιμετώπιση άλλων εταίρων. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε την ε, προσέγγιση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε με ε, το, στο δεύτερο γύρο των απαντήσεων με τον κύριο Σεάμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την κερδοσκοπία σχετικά με τις πρώτες ύλε γενικά, νομίζω ότι στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του G20 μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις βιομηχανικές ε, ε, πρώτες ύλες. Ε, όπως είπα πριν, οι χρηματοοικονομικές αγορές δεν διακρίνουν μεταξύ πρώτων υλών, αν είναι γεωργικές ή βιομηχανικές, αλλά εξαρτάται από, το είδος το οποίο θέλουν να επενδύσουν για να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους οι οικονομικοί φορείς. Δεν κάνουν λοιπόν διάκριση ανάλογα με το αν πρόκειται για ενεργειακές ή γεωργικές ή μεταλλευτικές πρώτες γιατί θα έχουμε περισσότερο διαρθρωμένο αντικείμενο εργασιών για τις γεωργικές και ενεργειακές πρωτεσίλες. Τις ενεργειακές πρωτεσίλες απλώς για να συνεχίσουμε αυτά τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν ήδη γίνει μέσα στο G20 και εμείς θα χτίσουμε πάνω σε αυτά. Για τις γεωργικές πρωτεσίλες ε, να το κάνουμε γιατί και αυτό υπάρχει ε, στα συμπεράσματα της ΕΟΥΛ, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Και οι προηγούμενες συνεδριάσεις του G20 δεν έδειξαν ότι υπάρχει ιδιαίτερη βούληση να υπάρχει μια διαρθρωμένη προσέγγιση για τις πρώτες ύλε από τον ε, ε, μεταλλευτικό και εξορυκτικό τομέα. Για, την, ε, για τον περιορισμό για τον περιορισμό των ανοιγμάτων στο χρηματιστήριο, ε, θέλω να πω ότι ως μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να χρησιμεύσει. Υπάρχουν κάποιοι τομεί που μέχρι τώρα δεν ήταν στην αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών και γι' αυτό μίλησα για τη διαφάνεια και είναι σημαντική η διαφάνεια Ξέρουμε τις ε, συναλλαγές που γίνονται έξω από, την, ε, από τα χρηματιστήρια και θέλουμε να αυξήσουμε τα μέτρα διαφάνειας ε, που υπάρχουν. Επίσης, πιστεύουμε στο συντονισμό μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών για τα προϊόντα αυτά καθεαυτά και για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία με ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στις αγορές εμπορευμάτων και στις αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα όταν θα χρειαστεί. Αλλά ως μέτρο ο περιορισμός των ανοιχτών θέσεων δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του μπορεί να μας καλύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεσά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να σχολιάσω για τη διαφάνεια. Νομίζω ότι είναι υψής της σημασίας το θέμα, διότι από το 2004 η αύξηση των, στις τιμές των αγαθών και οι διακοιμάνσεις στις τιμές, οι διαμάχες που συνεχώς γίνονται για τον έλεγχο των εισοδημάτων που προκύπτει από αυτές τις πρώτες ύλε, κάνουν τη διαφάνεια ένα απόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε πολιτικής για τα ορεικτά και από πλευράς εισαγωγών και από πλευράς εξαγωγών. Όπως είπε ο καθηγητής Πολ Κόλλιερ από την Οξφόρδη, η διαφάνεια θα έπρεπε να είναι το εφαλτήριο για οποιαδήποτε χώρα θέλει να κάνει είτε εισαγωγές είτε εξαγωγές. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό στις εξοριστικές βιομηχανίες. Έκανα μία σύμβαση, πέντε χώρες έχουν ε, επικυρώσει τους κανόνες, έγινε μία διάσκεψη στο Παρίσι το Μάρτιο και ε, πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα από πλευράς κοινωνίας των πολιτών ε, για τις χώρες που κύρωσαν ε, όλα αυτά, διότι πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία και συμφωνία, αλλά πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια ώστε να βελτιωθούν και οι συνθήκες ανάπτυξης των ε, ορυκτών υλικών, ε, πώς να βελτιώσουμε τις συμφωνίες που υπογράφονται από τις χώρες μας και πώς βελτιώνει τις ζωές μας, ε, ζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το βλέπουμε. Το θέμα λοιπόν της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει ολοένα και αυξανόμενη συνένεση μεταξύ των ε, χωρών ότι θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς ε, υπάρχουν βασικά ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πώς λαμβάνει μια κυβέρνηση από πλευράς ε, φορολογίας ε, για την ε, εξαγωγή αγαθών. Το βασικό ερώτημα είναι τι τα κάνει η κυβέρνηση αυτά τα χρήματα που παίρνει. Επίσης, ποιες διαδικασίες εντάσσονται στον προπολογισμό ώστε να ε, είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα κονδύλια δαπανώνται με τον κατάλληλο τρόπο. Και υπάρχει φυσικά και η άλλη άκρη του νομίσματος. Ε, αυτή τη στιγμή ε, γνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί αυτά τα κονδύλια. Ο πληθυσμός θέλει να μάθει τι γίνεται με τις συμβάσεις. Είναι σωστές οι συμβάσεις. Η χώρα έλαβε αυτά τα οποία δικαιούνται από τη σύμβαση ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία έκκληση σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ο ρόλος ε, των κοινοβουλίων ε, στις χώρες παραγωγούς ε, φυσικών πόρων είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει κάποιος τρόπος για να επεκτείνετε ίσως και εσείς την ε, συνεργασία σας με τα κοινοβούλια των χωρών που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους για να αυξήσουμε ε, τη διαφάνεια. Βέβαια η διαφάνεια δεν αρκεί εάν δεν είναι υπόλογη η κυβέρνηση για αυτά που γίνονται. Ο λαός δεν μπορεί να, ζητάει την να ρωτάει την κυβέρνηση γιατί έγινε κάτι και γιατί δεν έγινε κάτι καλύτερα εάν δεν είναι υπόλογη η κυβέρνηση για αυτά που κάνει. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ καλός κανόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να διδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις εταιρικέ σχέσεις και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ε, χωρών εταίρων τους για να βελτιωθούν οι γνώσεις τους στον τομέα τομέα και η διαφάνεια. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική πρόταση και την υποστηρίζω και εγώ να δημιουργηθούν εταιρικέ σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους και να προσπαθήσουμε να ε, γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χωρών εισαγωγέων και των χωρών εξαγωγέων και των επενδυτών και των χωρών που είναι πλούσιες σε πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά παράδοση ανάπτυξης γνώσης και τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς και θα μπορούσε αυτή η γνώση να ε, τεθεί στην υπηρεσία των χωρών αυτών για να βελτιωθούν οι εταιρικές σχέσεις αυτές και η συνεργασία και φυσικά να αυξηθεί η διαφάνεια και να υπάρχουν ε, συμμετρικά πληροφορίες. Αυτό είναι βασικό ε, για να απαντήσουμε στο ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα σήμερα και που σχετιζόταν με τις ε, παράνομες δραστηριότητες ε, για την ανάπτυξη των φυσικών πόρων, τη διαφθορά κατά την υπογραφή συμβάσεων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ισότιμη ε, μεταχείριση και ισότιμο πεδίο μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν. Αυτά αποτελεί τον ακρογωνια λίθο όλων όσων προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ καθηγητή Σέγκερτ για τον κύριο Κοφέρ που μου απίφθινε δύο ερωτήματα. Μπορώ να απαντήσω εν συντομία και στα δύο από αυτά. Καταρχήν, για τις ε, έρευνες που έκανε η κυβέρνηση Ομπάμα για τις ε, καταγγελόμενες ε, εμπορικές πρακτικές που αφορούν τον τομέα καθαρής ενέργειας στο... από την πλευρά των Κινέζων. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων για τα θέματα αυτά, μπορώ να σας δώσω ποια είναι η γενική μου, τη γενική μου εντύπωση. Νομίζω ότι η έρευνα αυτή για εμπορικές πρακτικές οι οποίες είναι αθέμητες ότι θα προσφύγει δηλαδή στον Παγκόσμιο Οργανισμό μπορεί αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σίγουρο. Νομίζω ότι πολλά για αυτό το περιεχόμενο αυτής της υποθέσεως εξαρτάται, εξαρτώνται από την ισορροπία μεταξύ δύο ζητημάτων <clears throat> από την, από την κινέζικη πλευρά επιχειρηματολογήσανε ότι οι περιορισμοί εξαγωγών οφείλονται σε προσπάθειες που κάνουν να βελτιώσουν την ε, περιβαλλοντική ποιότητα της εξόρυξης σπανίων γεών. Γνωρίζουμε πολλοί από εμά που είμαστε εκτός της Κίνας ότι δεν ακολουθούνται πρακτικές που θα το απαραίτητε στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Και η άλλη άποψη, αυτή δεν οδηγεί σε μια, αν το δούμε έτσι δεν είναι παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ, ενώ από την πλευρά των εργαζόμενων στη Χαλιβουργία που κατέθεσαν αυτήν την καταγγελία στις ΗΠΑ υπάρχει η άλλη άποψη του πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη που δίδεται από την Κίνα στους τομείς ε, που είναι εξαγωγικοί τομείς παραγωγής προϊόντων ε, καθαρής ενέργειας ότι οι περιορισμοί εξαγωγών είναι κυρίως μια κρυφή επιδότηση προς τον τομέα αυτό τον κοινωνιστικό και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αποχρόν λόγος για να προχωρήσει κανείς να ζητήσει την επίλυση διαφορών στα πλαίσια του ΠΟΕ. Επίσης μου ζητήσατε να σας εξηγήσω ποιες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με την νομοθεσία Dodd-Frank στις ΗΠΑ. Για αυτούς που δεν ξέρετε, πετύνος πρόκειται ακριβώς, είναι ένα μικρό τμήμα της ρύθμισης των του χρηματοπιστωτικού τομέα που τέθηκε σε εφαρμογή στις ΗΠΑ σε σχέση με ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων. Οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει τώρα να επαληθεύουν ότι οι εισαγωγές αυτών των ορυκτών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους δεν περιέχονται από περιοχές όπου σοβούν συγκρούσεις, ενόπλες συγκρούσεις και αυτό αφορά ιδίως το Ταντάλιο, στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό ή προσόδους από ορυκτά που ουσιαστικά τροφοδοτούν τους εμφύλους πολέμους και τις αναταρχίες, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής. Οι εταιρείε μας προσπαθούν, αγωνίζονται να εφαρμόσουν αυτούς τους νέους κανόνες. Η δική μου άποψη είναι ότι μια πλήρης εφαρμογή μπορεί να γίνει με κάποια χρονική υστέρηση γιατί οι περισσότερε εταιρείε προσπαθούν να καταλάβουν που προέρχεται. Προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Εταιρείε όπω η Apple και η Microsoft και άλλε, που ουσιαστικά είναι κατασκευαστέ των τελικών προϊόντων για τον καταναλωτή που περιέχουν τα ταντάλιο και άλλα προϊόντα από τέτοιε περιοχέ συγκρούσεων. Αλλά υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα βήματα στην αλυσίδα τροφοδοσία που χωρίζουν την εξόριξη του υλικού από την παραγωγή του τελικού προϊόντος και νομίζω ότι είναι σωστό να πει ότι εταιρείε όπως η Apple και η Microsoft δεν ξέρουν στην πραγματικότητα ποια είναι η τελική πηγή από την οποία προέρχονται τα υλικά που χρησιμοποιούν στου υπολογιστέ τους και προσπαθούν να βρουν ακριβώς από πού προέρχονται όλα αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο ερώτημα από τον κύριο Παραγιώτοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ο κύριος ε, κύριε Μπουτικόφερ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι ομιλητές. Σήμερα μπορέσετε <clears throat> να καταδείξετε όχι μονάχα το ενδιαφέρον που έχετε για την παγκόσμια κατάσταση σε σχέση με τους ε, φυσικούς αυτούς πόρους, αλλά έχετε παρουσιάσει και μια σειρά από προτάσεις για λύσεις. Και έχουμε δει πολύ καλά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Τώρα γιατί τα ονομάζω προβλήματα. Εγώ έχω ασχοληθεί με την ε, τεχνολογία εξόριξης ορυκτών εδώ και 30 χρόνια και εκπροσωπώ την Ευρώπη στο συνέδριο, στο συνέδριο, το Διεθνές Συνέδριο για τη μεταποίηση εξορισωμένων ουσιών. Υπάρχουν <clears throat> πρώτοι πρωτεσίλες και τέτοιοι πόροι αλλά πόσο κοστίζει στην Ευρώπη να αποκτήσει αυτούς τους πόρους για τη βιομηχανία της. Και το πρακτικό ερώτημα είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε τα 100-120 δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε σε διάφορες χώρες του κόσμου για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία μας έχει αυτά τα αυτούς τους, ε, τις πρώτες που τη βοηθούν να λειτουργήσει και την εξασφαλίζουν τη συνέχισή της. Καταρχήν για τους φυσικούς πόρους που μπορεί να εξευρεθούν στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι για οικονομικούς λόγους έχει μειωθεί η ε, δραστηριότητα στην Ευρώπη. Ήταν πολύ χαμηλές οι τιμές <clears throat> δεκαετία του 1990 και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση της εξορυκτικής βιομηχανίας. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλέ οι τιμέ. Ένα τόνο χαλκού κοστίζει 10.000 δολάρια. <clears throat> Θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ανακτηθεί η ικανότητα εξόρυξης. Αλλά παραμένουν και πολλά απόβλητα από την επεξεργασία ορυκτών για την απόκτηση μετάλλων. Αυτό αφορά την εξόρυξη χαλκού, μολύβδου, χρυσού πάρα πολλά μέταλλα. Λοιπόν, πώ θα αντιμετωπιστούν αυτά τα υπολείμματα. Όλα αυτά απαιτούν νέε τεχνολογίε, νέε μεθοδολογίε. Και στον τομέα αυτό μπορούμε πράγματι να επωφεληθούμε από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλή εμπειρία στα θέματα αυτά. Η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να επενδύσει σε αυτές τις τεχνολογίες και η Ευρώπη έχει την αντίστοιχη τεχνογνωσία. Έχω πάει σε εδώ σε όλες αυτές τις χώρες που έχουν τέτοιους φυσικούς πόρους που είναι έτοιμες να δώσουν και από τη δική τους πλευρά πόρους σε αντίτιμο της <clears throat> απόκτησης τεχνολογιών για αποδοτική χρήση της ενέργειας, διαχείριση υδατήρων πόρων κτλ. που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εν κατακλείδη νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές ευκαιρίες για συνεργασία γιατί κάποια μέταλλα μπορούν να ανακυκλώνονται στο διηνεκές. Αλλά ξέρουμε ότι η κατανάλωσή τους θα αυξηθεί στο μέλλον και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τη σωστή λύση η οποία θα εξασφαλίσει ότι έχουμε μια μακροχρόνια ασφάλεια τροφοδοσία σε πρώτε ύλε και στρατηγικά υλικά όχι μόνο για τι ΗΠΑ αλλά και για την Ευρώπη και όλε τι χώρε του κόσμου. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή τη συζήτηση γιατί ήταν πάρα πολύ καρποφόρα και χρήσιμη τουλάχιστον από τη δική μου προσωπική σκοπιά. Ευχαριστώ λοιπόν κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι έχετε μείνει τουλάχιστον. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλου του εμπειρογνώμονε μα, όχι μόνο για την παρουσία του και για τα ευφυή ε, επιχειρήματά μας που μας βοήθησαν να σκεφτούμε καλύτερα για το θέμα αυτό, αλλά για το γεγονός ότι προωθείτε όλοι προβληματικοί προβληματική για το θέμα αυτό. Υπάρχουν ακροάσεις όπου βγαίνει κανείς με μεγαλύτερη ανησυχία και περισσότερα ερωτήματα δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι μάθαμε πολλά πράγματα. Θέλω ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ και εξ του κυρίου Κόφερ ο οποίος είναι ο μας και ο οποίος έχει σταθεί ιδιαίτερα ενεργός στα θέματα αυτά. Παραμένει ακόμα ένα σημαντικό και δύσκολο εγχείρημα για μας, αλλά έχουμε πάρει πολύ, πολύτιμες πληροφορίες και μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα.